Right, everybody, we now have, have our... Τώρα είμαστε στην ώρα ψηφοφορίας. Πάρτε τις κάρτες σας και βάλτε τα στο μηχάνημα για να ελέγξουμε καταρχήν. Παρακαλώ. Um, right, we'll, we'll, we'll... Θα Κάνουμε ένα δοκιμαστικό πρώτα. Για να δούμε. Θα κάνουμε μυστική ψηφοφορία ή όχι. Όχι. Αν είναι μυστική μπορούμε να ελέγξουμε. Καλώς. Ωραία. Θα δούμε αν λειτουργεί η μυστική ψηφοφορία αν σας αρέσει ο διπλανός σας. Γι' αυτό ψηφίζουμε, λέει η Πρόεδρος. No, no, no, closed. No, no, no, because they still. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι? Όχι, από ό,τι βλέπω εγώ. Γι' αυτό παρακαλώ ψηφίστε Έχετε βάλει όλες τις κάρτες σας. Εδώ είναι πέντε που βλέπω ότι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Τέσσερις. Η Άστριντ, για παράδειγμα. Ωραία. Εντάξει. Όλοι ψηφίσανε και μάλιστα και ένας παραπάνω. Ή όχι. Όχι, εντάξει. Εντάξει είμαστε τώρα. 36 ε, λένε ότι τους αρέσει ο διπλανός τους. Τρεις όχι και τέσσερις αποχή. Ωραία. Οπότε περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες και πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε την έκθεση του Τέοτορ Δημήτρου Στόλογιαν για τις χρηματοπιστωτικές οντότητες υπέρ της τροπολογίας 1 κατά αποχές. Για να το λέξουμε, για να το λέξουμε, γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο. Πέρα στις ψηφοφορίες. Και τώρα είναι σαφές, με ενδιαφέρον. Τροπολογία 10 τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τζούρι 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, Α, μαζί την 11 μέχρι και τη 16. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται μαζί 18 με 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 89 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική β υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103. Όχι, καταπίπτει όπως και 104. Συμβιβαστική ε ή αγγλικό υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ μαζί η 31 μέχρι και 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά για να ελέγξουμε παρακαλώ την 112. Ψηφίστε. Δύο παραπάνω έχουν ψηφίσει στο ΕΛΚ. Τρεις παραπάνω. Τρεις λοιπόν πρέπει να βγάλουν τις κάρτες τους. Αναπληρωτές. Ναι. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καλά, να ελέγξουμε 113 γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Ψηφίσατε όλοι, πέρα τη προφορίες. Απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37 υπέρ, Δεν καταλαβαίνω καλά. Αποχές. Ψηφίζετε παρακαλώ γιατί δεν βλέπω καλά. 37. Θα ελέγξουμε γιατί δεν σας βλέπω καλά. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνετε. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μην ε, σηκώνετε το δάχτυλό σας, τα χέρια σας να σηκώνετε γιατί δεν βλέπω. 38 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική F, σίγμα τα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 Τι να ελέγξουμε. Voted, the vote. Πέρα στις προφορίες. Ε, είπα κι εγώ ότι εγκρίνεται και πράγματι. Από ό,τι φαίνεται εγκρίνεται. Δίκιο είχα. 128 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49. Με 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G, Z, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 55 με 57 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 με 64 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 134 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 65 με 76 μαζί και την τζούρι 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 135 τώρα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78. Με 83 μαζί και την 2 και 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 4 τώρα. Υπέρ,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 Με ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα θα ψηφίσουμε το τροποποιημένο κείμενο. Υπέρ παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 42 υπέρ και κανείς κατά. Και το νομοθετικό περιεχόμενο, το κείμενο νομοθετικού περιεχομένου παρακαλώ. Ψηφίστε παρακαλώ, ψηφίστε όλοι. Άλλοι δύο πρέπει να ψηφίσουν, άλλος ένας. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία, 43 υπέρ πάλι. Μπράβο, κανείς δεν είναι κατά. So actually, you have to read. Sorry for this. You have to read the same, but instead of credit default swaps, you say you say conglomerates. Otherwise, sorry. Right. Okay. Sorry about. Καλώς. Πρέπει να σας διαβάσω τώρα κάτι. Ψηφίσαμε μόλις τώρα την έκθεση για τις χρηματοπιστωτικές οντότητες. 20 χρηματοπιστωτικού ομίλου με πρόθεση να ξεκινήσουν ε, ε, διαβουλεύσει για πρώτη ανάγνωση. Είναι θέμα προς προτεραιότητα τη Επιτροπή μας. Βάσει των διαδικασιών η διαπραγματευτική εντολή είναι το σχέδιο έκθεση που μόλι ψηφίσαμε και η πρόεδρο, συγητή και σκιώδη συγητέ θα συμμετέχουν στην ομάδα διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχει αντίρρηση από ό,τι βλέπω. Αν έχετε, τώρα να μας το πείτε. Όχι, λοιπόν, δεν υπάρχει αντίρρηση. Συνεπώς, η διαδικασία θα προχωρήσει σε αυτή τη βάση. Εγκρίνει δηλαδή η Επιτροπή μας ότι προχωράμε σε προσπάθεια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Πάντα το κάναμε αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Προσπαθούμε τώρα, το κάνουμε και τυπικά. Περάμε τώρα στο σημείο 9 που είναι η ψηφοφορία Και άλλη ανακοίνωση πρέπει να σας κάνω σχετικά με τον κατάλογο ψηφοφοριών. Πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα θα είναι η τελευταία συνεδρίαση ΕΚΟΝ για την Σόνια Βουλνέι η οποία μετά από πολλά χρόνια δουλειά εδώ πηγαίνει στην μονάδα συναπόφασης από 1η Απριλίου. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο όλοι μαζί. Να εδώ είναι η απριλιου τις ευχομαστε οτι καλυτερο ολοι μαζι νατι εδω ειναι η σονια Σε ευχαριστούμε πολύ Σόνια. Θα φροντίσουμε να, το, να έχουμε και κάποιο ποτό. Τέλο δεν το ξέρει, αλλά κάτι θα τι οργανώσουμε. Περνάμε τώρα στο σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη, όπω έλεγα, που είναι η γνωμοδότηση και επιλογέ πολιτική για τη θέσπιση ενό ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για του καταναλωτέ και τι επιχειρήσει. Είναι η έκθεση του ΣΥΡΠΑ ποιητικά Είναι συμβαστική Α υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική γάμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δέλτα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε ή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Εδώ είχα τέσσερα διαφορετικά γκρι να διαλέξω. Τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο στο σύνολό του. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. 42 υπέρ και 2 κατά. Συγχαρητήρια, Σύρπα. So, now we're moving on to the... Τώρα περνάμε στους ορισμούς για τον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής με την σειρά Λιώπα και η Είναι μυστική ψηφοφορία αυτή. Θα ψηφίσετε συν αν είσαστε υπέρ του ορισμού και μείον αν είσαστε κατά. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα δούμε τελικά ποια θα είναι η σύστασή μας προς την Ολομέλεια. Υπέρ ή κατά. Βέρνερ. Ναι. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Για ποιον ψηφίζουμε. Έχουμε... έχουμε πρώτη Ναι, όπως είπα πρώτα η ΕΣΜΑ της Βερένα Ρος. Έσμα. Για την Βερένα Ρος. Αυτό ψηφίζουμε πρώτα. Μα υπάρχουν αρκετοί ψήφοι ΕΛΚ, θέλω να ξέρω. Υπάρχουν αρκετοί που ψηφίζουν ΕΛΚ, ναι. Α, εντάξει. Άμα είμαστε αρκετοί, ναι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 6 κατά και 4 αποχές. Η σύσταση μας θα είναι υπέρ του ορισμού αυτού. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία για τον Κάρλος Μοντάλβο, εκτελεσκός διευθυντής της ΕΙΟΠΑ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Δύο παραπάνω από το ΕΛΚ ψηφίζουν. Για βγάλετε δύο κάρτες. Οι αναπληρωτές. Ένας παραπάνω. Α, εντάξει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 4 κατά και 7 αποχές. Πάλι η σύστασή μας θα είναι υπέρ του ορισμού αυτού του κυρίου Κάρλος Μοντάλβο. Η τρίτη ψηφοφορία είναι για τον κύριο Άνταμ Φάρκα για την EBA. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Να αρχίσει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 38 υπέρ, 4 κατά και 3 αποχές. Και εδώ η σύστασή μας θα είναι υπέρ του ορισμού αυτού. Σας παρακαλώ, ε, έχουμε προτρέξει το χρόνο μας. Ο σκιώδης εισηγητής οι Περβόσπερες είναι στην Επιτροπή Επασχόλησης. Το κατανοώ αυτό βέβαια, είναι πολύ δύσκολο για τους πρόεδρους να έχουν διαφορετικές ε, προτάσεις. Έχουμε λοιπόν ένα τέταρτο διακοπή, πρωτού προχωρήσουμε στη συζήτηση του συστήματος αποζημίωσης επενδυτών. Right, thank you for that short interlude. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για αυτό το σύντομο διάλειμμα. Η ήρθε. Μπορεί λοιπόν να συνεχίσουμε με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε αρχικά προβλέψει. Περνάμε τώρα στην εξέταση των τροπολογιών για την οδηγία που αφορά τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών. Ο συγκεκριτής Όλη Σμιτ. Πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το θέμα έχει αναφερθεί στον τύπο λόγω πληρωμών στους ε, σεβουλευτές. Ε, λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτό και στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο εξετάζεται η υπόθεση αυτή. Ε, εν τω μεταξύ όμω ελέξαμε τι τροπολογίε και δεν υπάρχει καμία τροπολογία που έχει υποβληθεί από τα άτομα αυτά που κατηγορούνται στον τύπο. Και έτσι θα εξασθούν οπωσδήποτε όλε τι τροπολογίε από την Επιτροπή μα και θα εξεταστούν και θα συστηθούν όπω συνηθίζουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και τώρα να σα κάνω αυτή την δήλωση Πρόεδρου γιατί μου το ζήτησε και ο συγητής. Ουδέν νεότερο λοιπόν για την υπόθεση αυτή, αυτή τη στιγμή. Ζων Πολ, θέλετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν σκόπευα να μιλήσω για το θέμα αυτό που έχει ανοιχτεί προς το σύνολο του Κοινοβουλίου. Αν νομίζω είναι υποχρέωσή μας να ε, κάνουμε λίγη παιδαγωγική, γιατί διαβάζοντας την εφημερίδα έχω την εντύπωση ότι όταν ε, υποβληθεί μια τροπολογία έχει ήδη υιοθετηθεί και είναι στο κείμενο της οδηγίας. Είναι ασφαλμένο αυτό. Και από οικονομικής ε, πλευράς δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος θα πλήρωνε για να καταθεθεί απλώς μια τροπολογία. Αν έκαναν ότι τους κατηγορούνται οι βουλευτές αυτοί, είναι βέβαια αυτό πάρα πολύ κακό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει η ιδέα ότι δεν μπορεί κανένας να υποβάλει τροπολογίες ε, που να εμπνευστούν από κάτι. Εγώ σας το λέω ότι όταν μια τροπολογία είναι προς τη δική μου κατεύθυνση και είναι χρήσιμη, γιατί θα έλεγα ότι δεν είναι καλές. Θα πρέπει λοιπόν να το πω αυτό ξεκάθαρα. Να εξηγήσουμε ότι όταν μια τροπολογία περάσει από υποβληθεί μάλλον από το ένα βουλευτή θα περάσει καταρχήν από τους πολιτικούς φίλους του για να δει αν υπάρχει υποστήριξη. Μετά υπάρχει μια συλλογική εργασία για να ψηφιστεί ή να μην ψηφιστεί. Και δεν υπάρχει καμία άμεση σχέση ανάμεσα στην υποβολή μιας δραπολογίας και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Νομίζω ότι αν περάσουμε σε αυτό το λογικό θα έχουμε μια πολύ παράλογη θα πρέπει να προσπίσουμε νομίζω την ε, κοινοβουλευτική μας εργασία. Σε έξι χρόνια που είμαι εδώ, κανένα δεν μου πρότεινε να μου δώσει τίποτα για να υποβάλει κάποια τροπολογία. Αυτό είναι νομίζω μια πραγματικότητα. Εάν βέβαια κάποιο είναι απαταιώνα, ε, να τιμωρηθεί. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η εργασία μα. Και όσον αφορά τι τελικέ τροπολογίε που είναι συμβαστικέ τροπολογίε, αυτέ βέβαια προετοιμάζονται από το σύνολο των βουλευτών που ασχολούνται ε, με το θέμα, με τους ηγητές και τους κοιόδους ηγητές. Θα πρέπει νομίζω να το πούμε αυτό ξεκάθαρα για να μην δώσουμε λαβέ σε όλους τους αντιευρωπαίους και τους ε, που δρούν στον τομέα αυτό. Πρώτα σας ευχαριστώ, Ζαπόλ, έχετε βέβαια δίκιο και συμφωνώ μαζί σας. Μου φαίνεται ότι είναι κάπως σπατάλη χρημάτων να πληρωθεί κάποιος να υποβάλει μια τροπολογία. Και πρέπει να πούμε ότι πραγματικά τον υποβληθεί με τροπολογία, αυτό δεν αποκλεί κάποιε άλλες τροπολογίες. Καμιά φορά ίσως αυτό συμβαίνει. Σβέν, και συζητήσατε το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα. Και σας ευχαριστώ που λαμβάνετε το θέμα αυτό τόσο σοβαρά υπόψη και το διευκρινίσετε αυτό εδώ. Σας ευχαριστώ και για τα δικά σας σχόλια. Θα ήθελα να πω ότι ανησυχώ. Εάν κατάλαβα από τους τρεις κατηγορούμενους, ο ένας δεν έχει ακόμα παρατεθεί, παρετηθεί και εξακολουθεί να είναι ε, μέλος του σώματος. Έτσι καταλαβαίνω από τον τύπο. Είναι αλήθεια ή όχι. Επίσης ανησυχώ ότι εκείνος που θα αντικαταστήσει τον κύριο Στράσερ είχε επίσης μια εταιρεία λόμπι, είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του με έναν τρόπο που δεν θα έπρεπε να γίνεται ως ε, βουλευτής. Έχει διαγράψει βέβαια αυτή την, ε, την ιστοσελίδα, αλλά τα αντίγραφά της μπορεί να τα βρείτε στη δική μου, να το λάβετε υπόψη σας και να ζητήσετε από την πολιτική σας ομάδα να ελέγξει, να μην αντικαταστήσουμε κάποιον ε, μέλος του λόμπι με ένα άλλο μέλος του λόμπι. Πρώτα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα εξετάζεται από το αρμόδιο ε, αντιπρόεδρο, την Ταϊάννα Όλη, που είναι ω αντιπρόεδρο υπεύθυνη για την διαφάνεια και όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα τις τα υποβάλουμε και θα συνεχίσω να κρατώ τα μέλη τη επιτροπή εδώ ενήμερα για οποιοδήποτε αποτέλεσμα υπάρξει. Όπω σα είπα, εμεί ελέγχουμε όσο μπορούμε, αλλά όσον αφορά τι συγκεκριμένε τροπολογίε που συζητάμε αυτή τη στιγμή, όλα τα άλλα περνάνε από την Αντιπρόεδρο. Άστριτ. Ναι. Θα ήθελα να σας πω ότι αύριο θα εξετάσει το θέμα του Προεδρείου και θα πρέπει να περιμένουμε τις αποφάσεις του Προεδρείου της αύριο. Δεν χρειάζεται να το αναπτύξουμε εδώ και τώρα. Πρόεδρος, ναι, είναι σωστό αυτό. Γι' αυτό έκανα εγώ μία σύντομη ε, εισαγωγή, μια από αυτή η φάκελα αφορούσαν την εργασία της δικής μας Επιτροπής. Μπορούμε λοιπόν τώρα να θεωρήσουμε... ότι μπορώ να δώσω, το κλείσουμε το θέμα όσο το ξέρουμε εμείς και όλοι να πάρει το λόγο για να παρουσιάσει τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την σύντομη αυτή δήλωση. Ως εισηγητής είχα τρεις βασικούς στόχους στην έκθεση αυτή να αυξηθεί η προστασία του καταναλωτή για μεγαλύτερη κάλυψη, ανάγκη για καλύτερη εναρμόνιση των προγραμμάτων επένδυση στην Ένωση και τρίτον, βασικές αρχές για την αποζημίωση των επενδυτών. Υπάρχουν τέσσερα σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιαστούμε σήμερα. Το έχουν ε, ε, έχουμε πιο ευρύ το πλαίσιο Δεύτερον, ο χρηματοδοτικός μηχανισμός και οι αρχές. Τρίτον, το ύψος της αποζημίωσης. Και τέταρτο, ο μηχανισμός δανεισμού μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων. Το πεδίο. ισχύως. Επειδή υπάρχει ευρεία υποστήριξη, η αποζημίωση να καλύπτει και απάτες, ε, λειτουργικά λάθη όπως βλέπετε στις διάφορες τροπολογίες ή την 67 Ford, 68 της κυρίας Μπερές. Η κυρία Μπερές επίσης προτείνει σε κάποιες τροπολογίες της όπως την 56 όλες οι επενδυτικές εταιρείε να, κάνουν, να κλείνουν συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείε. Ενδιαφέρουσα η ιδέα αυτή αλλά θα αλλάξει εντελώ το σύστημα κατά τη γνώμη μου. Τολμηρή ιδέα. Ίσως η κυρία Μπερές καλό θα ήταν να μας ε, εξηγήσει λίγο παραπάνω το πνεύμα της τροπολογίας αυτής. Είμαι πέρα της ασφάλισης και εγγύηση για τις συσφορές ε, στο τρέχον σύστημα να εισαχθεί σε προαιρετική βάση θα μπορούσαμε να το προτείνουμε στην Κομισιό να κάνει μια μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων και μετά να μας προτείνει στο Κοινοβούλιο να εισάγουμε αυτό το προαιρετικό σύστημα. Η κυρία Μπέρες επίσης θέλει να πει ε, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι τοπικές αρχές να μπουν και αυτές οι 22 και 61. Όλες οι υπηρεσίες επενδύσεων υπό το MIFID και όλες οι δραστηριότητες πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία αυτή ICS. Εγώ θεωρώ ότι οι προτάσεις αυτές καλύπτονται από τις αλλαγές. Και μετά ένα καυτό θέμα, δύσκολο, συμπερίληψη των usage. Υπάρχουν μερικές τροπολογίες και για τα usage. Δεύτερον, το ύψο τη αποζημίωση Συμφωνώ με την Κομισιόν ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση, για την, ε, πλήρης ε, αποζημίωση για την, στην εναρμόνιση, έτσι να υπάρχει επαρκή και παρόμοια προστασία σε όλες τις χώρες της Ένωσης, γιατί τα προβλήματα που ζήσαμε τα ξέρουμε. Και βλέποντας τις τροπολογίες, θεωρώ ότι σήμερα υπάρχει πλειοψηφία υπέρ του να αυξηθεί το επίπεδο της αποζημίωσης από 50.000 ευρώ που προτείνει η Κομισιόν στα 100.000 ευρώ. Τροπολογία 81 της κυρίας Μπερές και 82 του κυρίου Κλούτε. Είμαι υπέρ των τροπολογιών αυτών. Τρίτον, ο χρηματοδοτικός μηχανισμός, funding mechanism. Ε, η Κομισιόν προτείνει ένα εκ των προτέρων, προτέρων χρηματοδότηση. Οι Βρετανοί συνάδελφοι, η Βίκη Φόρντ και εσείς, κυρία Πρόεδρε, είστε υπέρ ενός συνδυασμού χρηματοδότησης εκ των προτέρων εκ των υστέρων. Στην περίπτωση Φίνιξ, στη Γερμανία είδαμε ότι υπάρχει ανάγκη για χρηματοδότηση εκ των προτέρων και είναι δύσκολο να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ χρηματοδότηση εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Είμαι κατά των τροπολογιών αυτών. Για συζήτηση φυσικά είμαι στη διάθεσή σας και φυσικά θα γίνει και συζήτηση και στο Συμβούλιο. Το κόστος χρηματοδότησης θα το φέρει ο επενδυτής. Γι' αυτό πρέπει να είναι σε αναλογικό επίπεδο για τον επενδυτή. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ μιλάμε για βάρος, για άχθος, για τον επενδυτή και για όλο τον κλάδο. Πήγα στην Αθήνα πρόσφατα, είχα μια συνάντηση και συνάντησα και υπουργού και προσώπους από τον κλάδο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι ανησυχούν βάζουμε επιπλέον απαιτήσει και βάρη στις επιχειρήσεις και είναι δύσκολο να βγούνε έτσι από την ύφεση. Εγώ προτείνω 0,3% καταθέσεις στην πρότασή μου. Τα μέλη του ΕΛΚΑ, όπως η συνάδελφος Άλμπα, στην τροπολογία 100 προτείνω να μειωθεί από το 0,5% στο 0,1% η εισφορά. Και αυτό προς συζήτηση. Είπα και πριν ότι πρέπει να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία και να ξέρουμε τι κάνουμε όταν επιβάλλουμε τέτοιου είδους εισφορές. Τέσσερα, ο μηχανισμός δανεισμού. Ο προτινόμενος μηχανισμός είναι μηχανισμός αγγελεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Άρα είναι θετικός ως μέτρο. Η τροπολογία 144 Μπερές διαγράφει το μηχανισμό αυτόν και προτείνει ένα ευρωπαϊκό ταμείο από το οποίο να μπορούν να δανείζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό έχει σχέση με αυτό που είπα πριν. η συνάδελφος Μπερέση θα πρέπει να μας το αναλύσει λίγο. Δηλαδή κάθε εταιρεία να δίνει 5% από τα ασφάλιστρα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ασφάλισης με ανησυχεί λίγο αυτό. Τι, τι, τι θα είναι αυτό το τεράστιο ταμείο και πώς θα λειτουργεί, δεν ξέρω. Ο κύριο Άλμπα, 136, λέει τα κράτη-μέλη να μπορούν να δανείζονται το ένα από το άλλο μετά από 10 χρόνια. Εγώ η πρόταση εδώ είναι 5 χρόνια. Τέλος, είμαι υπέρ ορισμένων τροπολογιών του συνδέφου Γκίγκολτ, την 107 και την 108, και την 158 και τελειώνω με το εξή. Με την άριστη ομάδα στη γραμματεία μας, στην επιτροπή μας, και με τη δική μου επιδεξιότητα και βοήθεια βέβαια, και από κοινού και με την Ουγγρική Προεδρία και φυσικά με την Κομισιόν, όλοι μας προσπαθήσαμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις και θα το συνεχίσουμε αυτό και τις επόμενες εβδομάδες. Μερικοί μπορεί να θεωρείτε. ότι είμαι ένας φιλελεύθερος ο οποίος συνεχώς βάζω στο μάτι όλο τον κόσμο. Μερικές φορές είναι, είναι λογική αυτή η κίνηση. και θεωρώ ότι τμήμα του, της φιλοσοφίας του φιλελευθερισμού είναι να είναι κανείς λογικός και νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε. Ίσως το κύρια προβλήματά μας δεν είναι εδώ, στην δική μας στην Επιτροπή, τα προβλήματα ούτε στην Κομισιόν, κάπου αλλού είναι. Καλύτερα να μην πω πού μπορεί να βρίσκονται τα προβλήματα. Πιστεύω πάντως ότι θα καταλήξουμε σε καλή έκθεση και ελπίζω να έχω ευρεία υποστήριξη. Η δουλειά ήδη ξεκίνησε και θα έχετε και πλέον στοιχεία όπως θα περνάνε οι μέρες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πάμπλο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την ε, διαθεσιμότητά του και για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Έτσι κι αλλιώς είναι απόλυτα λογικός, οπότε δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα απολύτως. Συμφωνούμε σε πάρα πολλά σημεία με τον εισηγητή, περίπου σε όλα. Συμφωνώ με την πρότασή του να μην συμπεριλάβουμε τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα usage, και υπάρχει εξάλλου μία οδηγία για τους οργανισμούς αυτούς και υπάρχει και μία αναθεώρηση για τον οργανισμό αυτόν και αν ε, δεν καλύπτει απόλυτα τους οργανισμούς αυτούς, τότε μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά δεν έχει νόημα τώρα να συμπεριλάβουμε τους οργανισμούς αυτούς στην οδηγία που ετοιμάζουμε. Όσον αφορά για το επίπεδο κάλυψης, συμφωνούμε να αυξηθεί στα 1000 ευρώ. Πρέπει εξάλλου να πάμε σε περισσότερη αναρμόνιση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όσο νομοθετικά προχωράμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εναρμονίζουμε και τα κριτήρια τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα ακόμα. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούμε να ζητάμε από ορισμένε χώρες να μειώσουν την κάλυψή τους, άρα πρέπει να αυξηθεί αλλού και να υπάρξει εναρμόνιση στα 1000 ευρώ της κάλυψη αυτή, όπω λέει και ο έτσι και εγώ προτείνω να μειωθεί στο 0,1% η χρηματοδότηση των ε, ενεργών που καλύπτονται. Είναι ένα ποσό λογικό κατά τη γνώμη μας, μια που είναι κάτι που χρησιμοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις μόνο. Γι' αυτό και πιστεύουμε, ο μηχανισμός αυτός, γι' αυτό και πιστεύουμε ότι το 0,1% είναι ικανοποιητικό επίπεδο. Έρχομαι τώρα στις προθεσμίες. Προτείνω να παραμείνουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 10 έτη δηλαδή για την χρηματοδότηση του συστήματος. Την κάλυψη την ε, αλλάζουμε σημαντικά, οπότε νομίζω ότι τα 10 χρόνια είναι ένα καλό χρονικό διάστημα όσον αφορά τώρα τα εθνικά δάνεια. Και εδώ συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή. Η πρόταση της Επιτροπής πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, προς την αναρμόνιση και συμφωνούμε με αυτό, αλλά συμφωνώ με τον εισηγητή για το ότι πρέπει να περιορίζεται στο 5% και ότι το σύστημα δανείων μεταξύ χωρών δεν πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί παρά μόνο εφόσον έχει υπάρξει χρηματοδότηση του 100% των συστημάτων αυτών. Για να αποφύγουμε κίνδυνο για free riders. Έπειτα έχουμε και μια τροπολογία η οποία λέει ότι ο μηχανισμός αυτός δεν πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί παρά μόνο εφόσον υπάρχουν νομικά οι αναγκαίες εγγύσεις ότι οι πληρωμές ε, θα ε, λαμβάνονται χωρίς καμία δυσκολία. Θα υπάρξει αποκατάσταση πλήρης. Όσον αφορά τώρα για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, θέλουμε μια διευκρίνηση ότι οι επενδύσεις οι οποίες συνδέονται με την χρηματοδότηση άμεσα ή έμεσα τρομοκρατικών ομάδων δεν θα μπορούν με τίποτα να αποζημιωθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για περιφέρειες και χώρες όπως είναι η δικιά μου, όπου υποφέρουμε από τη μάστιγα της τρομοκρατίας. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή και εσάς κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Υπερβάνση τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα τηρήσω κι εγώ το ωράριο. Σας ευχαριστώ που τηρήσετε το ωράριο εργασιών μας όπως είχε προβλεφθεί. Πριν κάνω την εναλλακτική πρόταση που τη χαρακτήρισε θαραλέα ο εισηγητής. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το όλο περιραίους ατμόσφαιρα του κειμένου αυτού. Από τη μία μεριά έχουμε τα μύφ, από την άλλη μεριά έχουμε τα usage, το κείμενο αυτό και το κείμενο για τις ε, καταθέσεις και τις τραπεζικές εγγύησεις. Και τρέχουμε συνεχώς πίσω από τις χρηματοπιστωτικές αγορές προσπαθώντας να βρούμε ε, κάτι που να μην αποτελεί ανακολουθία, που να σέβεται το κείμενα και να επιτρέπει να κάνουμε γέφυρες μεταξύ των διαφόρων κειμένων και γράφων, που είναι ο εφιάλτης του νομοθέτη. Μια από τις μεγάλες δυσκολίες για το κείμενο αυτό εδώ είναι το ότι να δούμε πώς εναρμονίζουμε το ποσό των εγγυημένων ποσών με το κείμενο για τις καταθέσεις και ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί το συζητήσαμε πριν κάνει την έκθεσή του και έλαβε υπόψη τα σχόλιά μας και πρότεινε να ανέβουμε σε 100.000 γιατί εγγυημένα κονδύλια, ποσά μάλλον, έτσι ώστε να είναι ελεύθερος ο καταθέτης και να διαλέξει θα είναι καταθέσεις, η μορφή που θα έχει τα χρήματά του ή με άλλο τρόπο. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή που το δέχτηκε αυτό. Τώρα για τα κείμενο για το usage. Το πεδίο εφαρμογής του κειμένου αυτού βλέπουμε ότι υπάρχει μια πραγματική δυσκολία. Γιατί υπάρχει, αν υπάρχει ένα επενδυτικό προϊόν για το οποίο ε, οι ιδιώτες μένουν στην Ένωση είναι ακριβώς αυτά. Τα usage και κάνουμε ένα κείμενο για να εγγυηθούμε όχι μόνο τις επενδύσεις, αλλά δηλαδή για την κακή συμβουλή, λαθροχειρίες κλπ. Και το αποκλείουμε, αυτό που λέμε στα γαλλικά, ευέμ. Ε Ή τα αφήνουμε αυτά για κάποιον άλλο, για μια πράξη χώρισης όπως λέει ο κύριος Γκίγκολ, για μετά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας που αφήνουμε. Γιατί δεν είναι παράλογο να κάνουμε μια πρόταση σε σχέση με αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Διότι τι μας προτείνει η Κομισιόν. Μας προτείνει να έχουμε αυτό το σύστημα εξάντε εκ των προτέρων. Ενοχλεί τους Βρετανούς και άλλες αντιπροσωπείες, ούτε η κυρία Λούγιν της πολύ αρέσει το σύστημα αυτό. Και μας λέτε για το πεδίο εφαρμογή περιμένετε τα usage. Εγώ να περιμένω. Δεν πιστεύω όμως ότι η Κομισιόν θα βγάλει πρόταση μέχρι τον Ιούλιο γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε το χρόνο από σήμερα μέχρι τον Ιούλιο για να μελετήσουμε την βιωσιμότητα της πρότασης που κάνω εγώ. Συν 27 τροπολογίες, γιατί έχω καταθέσει πολλές. 27 τροπολογίες σχετίζονται με το θέμα αυτό. Να έχουμε ένα σύστημα ασφάλισης. Που σημαίνει αυτοί που προσφέρουν στο κοινό στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογή του ΜΥΦΙΤΣ και θα αναφερθώ αυτό σε λίγο. Επενδυτικά προϊόντα που ξαφνικά αποτελούν αντικείμενο λαθροχειριών κλπ. Εμπίπτουν επασφαιρτό σε πεδίο εφαρμογή τη οδηγία να καλύπτονται από έναν μηχανισμό ασφάλιση. Θα είναι χρήσιμο για την οικονομία και δεν θα έχουμε τις συζητήσεις που είχαμε ποιος εκ των προτέρων, εκ των υστέρων, τι και αλληλεγγύη μεταξύ των μηχανισμών αν υπάρχει ασφάλιση, να υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασφάλισης που ανάλογα με τα ασφάλιστρα θα πληρώνει. Άρα έτσι υλοποιείται αυτή η πρόταση. Τώρα για τα άλλα τα οποία ανάφερε ο συγητής για να μην σας φάλω χρόνο. Ξέρω ότι αποκλίνει από την αρχική πρόταση της Κομισιόν και θα μου πείτε «Α, ναι, ας ευχαριστήσουμε την Ουγγρική Προεδρία κλπ». Ε, θα εγώ, τι γίνεται με τα usage και γιατί να περιμένουμε μέχρι τότε. Δύο λόγια ακόμα για το πεδίο εφαρμογής. Ο εισηγητής είπε ότι έχει το αυτή το ανοιχτό να ακούσει, ενδεχομένως να ενσωματώσει στο κείμενό του το θέμα της bad advice που υπάρχει στην Αγγλία και το βλέπουμε και στο MIF. Νομίζω αξίζει αυτό να μπει στην οδηγία ως, όσον αφορά τις μικροοντότητες, μικροαντιτέ, τις τοπικές αρχές και τις μικροδοσκοπικές οργανώσεις που ανάφερα. Αν δούμε τον ορισμό του μυφ, κύριε Σιγητά, δυστυχώς δεν καλύπτονται αυτοί οι άλλοι που αναφέρατε από την εμπειρία που είχαμε όταν ξεκίνησε η κρίση. Τουλάχιστον στη Γαλλία, ίσως και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία λέει, υπήρχαν πολλές τοπικές αρχές οι οποίες αποσταθεροποιήθηκαν και είχαν ανάγκη να ισχύει και για αυτούς η εγγύηση για τις καταθέσεις. πρέπει και αυτοί να καλύπτονται από την κακοδιαχείριση στα πλαίσια των επενδύσεων που κάνανε. Το ύψος της αποζημίωσης, το ποσό μάλλον, που θα πρέπει να προεισπράτεται τα ασφάλιστρα, θα, ε, ο όρος θα επέτρεπε να καλύψουμε το 5% που ζητάνε μερικοί, 3% που ζητάνε άλλοι και 1% που ζητάνε κάποια άλλη τρίτη. Αυτά είχα κυρία Πρόεδρε να πω αυτή τη στιγμή λαμβάνοντας υπόψη ότι ουσιαστικά η, η πρόταση αυτή είναι μια εναλλακτική πρόταση αλλά θέλω να έχουμε το θάρρος στο Κοινοβούλιο να ζητάμε από την Κομισιόν να μας μελετάει χωρίς να μας λέει ότι έχουν προχωρήσει τα πράγματα ήδη Όντω έχει ξεκινήσει αυτή η υπόθεση εδώ και χρόνια. Πολλές τροπολογίες μας λένε ισχύσει μετά από 10 χρόνια πλήρω. Είναι πιο λογικό να περιμένουμε την αναθεώρηση των usage. Άρα να περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι. Σαΐντ. Ευχαριστώ πολύ που υπενθυμίζετε ότι η δικιά μου ομάδα είναι μεγαλύτερη. Μερικές φορές παίζει ρόλο. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για την δουλειά τους. Η συζήτηση αυτή δείχνει ότι όντως θέλουμε κάτι να πετύχουμε σημαντικό, ότι θέλουμε οι επενδυτές να έχουν εμπιστοσύνη στα προϊόντα στα οποία επενδύουν. Ορθό αυτό. Εκεί που διαφωνώ εγώ με κάποιες από τις τροπολογίες είναι στο θέμα της ηθικής ζημίας Ζητάμε δηλαδή να είναι προσεκτικοί οι επενδυτές και να λαμβάνουν την ευθύνη όταν επενδύουν. Εγώ λοιπόν, όταν υπάρχει κατάχρηση, κακοδιαχείριση, σε τι επίπεδο όμως. Πότε μιλάμε για κακοδιαχείριση. Κάποιοι επενδυτές που ακολουθούν διαφορετικά μοντέλα επενδύσεων μπορεί να ξέρουν ότι επενδύουν σε χώρες ή σε προϊόντα όπου να υπάρξει διαφορετική κάλυψη από αυτές την οποία είναι συνηθισμένοι, αλλά είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυτό το κίνδυνο και να κάνουν αυτή την επένδυση, επειδή αν πάει καλά θα έχουν υψηλά κέρδη. Να προστατεύουμε τους επενδυτές που δεν είναι καλά ενημερωμένοι, αλλά όχι και αυτούς οι οποίοι είναι καλά ενημερωμένοι και θέλουν παρόλα αυτά να επενδύσουν. Η διαφάνεια είναι κάτι που συζητάμε πολύ και θέλουμε και γι' αυτό το ζητάω και εγώ με τη δικιά μου την τροπολογία. Να υπάρχει διαφάνεια ώστε οι επενδυτές να ξέρουν τι πληρώνουν και τι κέρδος θα έχουν. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς λοιπόν και να δούμε σοβαρά την ιδέα μιας ε, ασφάλισης. Δεν λέω ότι πρέπει να έχουμε μαζικά συστήματα και να δεσμεύονται χρήματα σε αυτά. Όχι, αλλά όλοι θέλουμε την ιδέα της ασφάλισης. Η βασική μου ιδέα είναι η διαφάνεια και να ξέρουν για αντισταθμιστικά συστήματα τι πληρώνουν οι επενδυτές. Και κάθε φορά που προσθέτουμε ένα κόστος, το πληρώνει ο επενδυτής. Άρα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μια ισορροπία. Γιατί μερικέ φορέ οι επενδυτέ θέλουν να πληρώσουν αυτό το κόστο, αν υπάρχει ασφάλιση δηλαδή, είναι διατεθειμένοι να την πάρουν, θέλουν να έχουν τη δυνατότητα. Αλλά από 20.000 ε, pounds για το Λονδίνο, για τους επενδυτές στο Λονδίνο, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά φαντάζομαι ότι άλλοι επενδυτές σε πιο μικρές ή σε πιο καινούριε χώρες μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 20.000 pounds είναι πολύ για αυτούς. Και δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει για τις δικές τους χρηματοπιστωτικές αγορές. Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι το Λονδίνο και να πω πάρα πολύ ωραία. σε σύγκριση με μένα όλοι οι άλλοι μπορεί να ακούγονται σοσιαλιστές. Πάντως εγώ θα ήθελα ένα πραγματικό ανταγωνισμό και θέλω και τις μικρές ε, και μεσές ε, χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να τις δω στο Λονδίνο. Και συμμερίζομαι την άποψή σας ότι δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε εδώ ναι, τους ε, ΟΣΕΚΑ, έτσι, τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, τα USAGE. Μην έχουμε διπλές και τριπλές ρυθμίσεις. Όταν βλέπουμε την αναθεώρηση για τα usage, για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, πρέπει να καθησυχάζουμε ανησυχίες. Κυρίως για το Μέντοφ. Είμαι υπέρ της ε, ελεύθερης διαχείρισης, είπαμε να μην πληρώνουν τα πάντα οι επενδυτές, όμως τι χρήματα πρέπει να βάλουμε στα συστήματα αυτά. 0,5% λέει η Επιτροπή, 0,3% λέει ο συγγετής. Από πού θα τα βρούμε αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα το 0,3% θα το προτιμήσουμε επειδή είναι λιγότερο από το 0,5% αλλά παραπάνω από το 0,1%. Ε, από πού θα τα βρούμε αυτά τα χρήματα μην πετάμε νούμερα δεξιά και αριστερά χωρί να ξέρουμε σε τι ανταποκρίνονται ακριβώς, για να ξέρουμε και ποιο είναι το καλύτερο νούμερο τελικά. Δεν θα ήταν καλύτερα τα χρήματα αυτά να κυκλοφορούν στις οικονομίες μας αντί να κάθονται κάπου δεσμευμένα. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό σε βάθο για να δούμε ποιο θα είναι το σωστό ποσό ποσοστό πιο σωστά. Ευχαριστώ πάντως και τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, πρέπει να τη σκεφτούμε περισσότερο αυτή την οδηγία, αλλά εγώ ευχαρίστω θα συνεχίσω τη συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις. Ευχαριστούμε. Σβέν. first, thanks a lot uh, to... Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον σοσιαλιστή φιλελεύθερο εισηγητή και όλους τους συναδέρφους Πάντα είχαμε καλές επαφές και συναντήσεις και υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο σύγκλησης. Το βασικό είναι ναι στον ανταγωνισμό, αλλά όχι σε ανταγωνισμό που να βασίζεται σε αποφάσεις που αναγκάζονται να παίρνουν οι επενδυτές όταν δεν γνωρίζουν ποια είναι ακριβώς η κατάσταση, οπότε κινδυνεύουν να είναι θύματα καταχρήσεων και απατών. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν αυτά τα συστήματα εγγύσεων. Το ερώτημα που τίθεται για μένα και που έθεσε και η Περβάνς είναι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλιση, αυτή να είναι η λύση. Αμφιβάλλω για το κατά πόσο κάτι τέτοιο θα ήταν ευθυνότερο, θα ήταν ευθυνότερη λύση. Ιδεολογικά δεν έχω άποψη γι' αυτό. Δεν είναι ιδεολογικό το θέμα. Έχει νόημα να βρούμε μια λύση για να προστατεύσουμε τους επενδυτές με το φθηνότερο δυνατό τρόπο από απάτες και καταχρήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λύση. Μια ιδιωτική αγορά δεν είναι πάντα η πιο φτηνή, η πιο φτηνή από μια συνεταιριστική λύση, γι' αυτό και με εκπλήσει λίγο αυτό που άκουσα. Επιμένω, δεν είναι ιδεολογικό το θέμα για μένα. Είναι το ποια είναι τελικά η πιο φτηνή λύση. Γιατί τα χρήματα στο τέλος που χάνονται, από, το, από τα έσοδα που δημιουργούν οι επενδυτές. Εμείς δεν θέλουμε την πιο ακριβή αγορά, θέλουμε μια φτηνή λύση ώστε ο ανταγωνισμός να λαμβάνει χώρα εκεί που θέλουμε να λαμβάνει χώρα. Σε επίπεδο δηλαδή των, των διάφορων φορέων οι οποίοι βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους για να τραβήξουν τις ε, αποταμιεύσεις. Παρατηρήσεις τώρα για το επίπεδο. Είναι θέμα υπολογισμού. Πάλι δεν είναι θέμα πολιτικών διαπραγματεύσεων και παζαριών. Συμφωνώ με αυτό. Για τους ΟΣΕΚΑ, τα usage. Είναι ένα από τα πιο βασικά ζητήματα. Το λόμπι το μεγαλύτερο που έγινε ήταν για τους οργανισμούς ακριβώς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Μην επαναλάβω τα ίδια επιχειρήματα. Είναι βασικό ότι περιπτώσεις όπως είναι της Μέντοφ πρέπει να χαίρουν προστασίας. Ο κίνδυνος είναι σχετικά χαμηλός, γιατί είναι ένας ρυθμισμένος τομέας, βέβαια όχι και πλήρως, πρέπει να υπάρχει συνεπώς μια προστασία. Αν έχουμε τη στήριξη όλων των πολιτικών ομάδων, μπορούμε να το δούμε αυτό όταν κάνουμε την αναθεώρηση για τους ΟΣΕΚΑ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί που έκαναν λόμπι εδώ θέλουν να αποκλειστούν. Δεν υποφελείται ο καταναλωτής, το αντίθετο είναι. Γι' αυτό θα ήθελα εδώ να καταλάβω καλύτερα από τους συναδέρφους τι θέλουν. Θέλετε να πάει το θέμα αυτό στην αναθεώρηση των ΟΣΕΚΑ ή θα στηρίξετε να υπάρχει μια εγγύηση στα πλαίσια των ΟΣΕΚΑ, οπότε να προστατευτούν και οι καταναλωτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως όλους για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Ευχαριστώ και τους πράσινους που μας οδήγησαν σε αυτή την τοποθέτηση και ελπίζω ότι θα βρούμε κάποια λύση. Για την λύση ασφάλισης της Περβάνς, πάντως είναι κάτι που πρέπει να δούμε σε βάθος σε άλλη συζήτηση που θα κάνουμε μεταξύ μας οι σκιώδεις και όποιος άλλος ενδιαφέρεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γιώργα. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Ε, Jean Paul. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσει. Πρώτον, νομίζω ότι το θέμα των ασφαλίσεων αξίζει να μελετηθεί. Όχι μόνο εν παρόδο, είναι μια λύση ενδιαφέρουσα, γιατί όπως είπε και η κυρία Μπερέτς, θα μας επιτρέψει να παραμείνουν τα ποσά αυτά μέσα στην οικονομία, να μην τα εξοδοτερώσουμε. Και δεύτερη παρέστηση, όσον αφορά τα ΟΣΕΚΑ, τα USITS, πάντα άσχημο είναι να βιαζόμαστε υπερβολικά. Εκτός αυτού, μία καθυστέρηση μερικών μηνών δεν θα ήταν και πάρα πολύ ενοχλητικό θέμα. Εδώ το φάκελο που με απασχολεί, που ολοκληρώνεται το 2018, Μπορούμε να σπαταλήσουμε κάποιους μήνες. Και αυτό θα πρέπει νομίζω να έχουμε κατά νου και όχι ε, κάθε φορά να λέμε ε, θα το δούμε σε μερικού μήνε, αλλά έπρεπε να το έχουν κάνει πιο πριν και λοιπά. Ας είμαστε κάποιο πιο λογικοί και συνεπείς Και με μερικούς μήνες καθυστέρηση δεν πειράζει καθόλου λόγω του ρυθμού στον οποίο ζούμε. Θα ήθελα να ήταν πιο γλίγορα, αλλά πρέπει να συμμορφώ με την πραγματικότητα. Αυτές οι προτάσει της ε, κυρίας θα πρέπει να μελετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για Άστριτ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Χωρί να επισέλθω σε λεπτομέρειε, θα ήθελα να αναφερθώ σε γενικές γραμμές της τροπολογίες που υπέβαλα για την έκθεση αυτή. Είχα και την ευκαιρία να τη... Δεν είχα ακόμα την ευκαιρία να τη ε, κουβεντιάσω με τον κύριο Σμιτ. Έχω την ε, εντύπωση ότι δεν είναι τελείως ανώδυνες αυτές οι τροπολογίες. Το να εξορίσετε το 0,5 ω 0,1% ίσως σας φαίνεται πολύ απότομο, αλλά αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε στα πλαίσια οδηγίας αυτής για πολύ σπάνιες και μεμονωμένες περιπτώσεις. Βέβαια, πρέπει να προβλέψουμε ε, πόρους εγγύησης γνωρίζοντας ότι ε, οι αποζημιώσεις θα χρειαστεί να γίνουν σε πολύ ακραίες περιπτώσεις. Υπό τους όρους αυτούς, ε, μία συμβολή, αν μπορώ να την πω έτσι, της τάξης του 0,5% δεν είναι καθόλου ρεαλιστική. Θα πρέπει λοιπόν να το επανεξετάσουμε το σημείο αυτό και να μειώσουμε το ποσοστό. Όσον αφορά τη λήψη υπόπτων σε μέσα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή. Πολύ καλά τα είπε και η κυρία Μπερές. Ε, εκείνο, εκεί που δεν συμφωνώ μαζί της είναι ότι η οδηγία ΟΥΣΕΙΤΣ 5 θα τεθεί στην ημερήσια διάταξη και η ευθεία της καταθέτουσας ε, τράπεζας θα πρέπει να διευκρινιστεί άποψη διαπαντός. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση προτού σκεφτούμε να συμπεριληφθούν τα, τα, τα υπόρρια αυτοί στην ευέλα της εν λόγω οδηγίας. Τούτων εχθόντων, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, κυρία Πρόεδρε, θα μπορούσε να τα χρήσιμο πλήρως μόνο εάν οι ευθύνες κάθε είναι απόλυτα ξεκάθαρες και δεν υπάρχουν επικαλύψεις ή ασάφειες που πρέπει να απεφευχθούν πάθηση θυσία. όπως το είπε και ο κεφαλής μου ο κ. Γκοζές, είναι επίγον να περιμένουμε. Όσον αφορά τώρα τις αποζημιώσεις, τις οποίες θα είχαν δικαίωμα οι επενδυτές, μου φαίνεται το εξή πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε απόλυτη εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω. Η εγκαθίδρυση ελαχίστου κατοφλίου μου φαίνεται ότι θα ήταν η καλύτερη των λύσεων. Εγώ πρότεινα 50.000, άλλοι συνάδελφοι θέλουν 30.000. Να το συζητήσουμε το θέμα. Κάνω να το ολοκληρώσω. Μία τελευταία παρατήρηση για τη μεταβατική περίοδο. Είναι σαφές ότι η υποβολή των πόρων αυτών εκ των προτέρων εξάντε δεν θα είναι και πολύ γλίγορο ή εύκολο. Και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου η διάρκεια της μεταβατικής περιόδους περίοδου θα εξαρτάται από τις απαιτήσει που θα επιβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί όσο πιο αυστηρές είναι οι προδιαγραφές αυτές τόσο πιο πολύ χρόνο θα πρέπει να δώσουμε στον τομέα. Αν ζητήσουμε κάτι το αλαφρό, μπορούμε να ζητήσουμε μια θέση ισχύ πιο γρήγορη. Ας το έχουμε αυτό απόλυτα κατά νου. Και όπως είπε ο κ. Κροζές, ζήτω η λογική και συνοχή στον τομέα. Ευχαριστώ. you. Mr. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και τους Κιώδης για τη δουλειά τους, λέει ο κύριος Φέιο. Και θέλω να κάνω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, το σύστημα ασφάλισης. Νομίζω ότι πρέπει να μελετήσουμε το θέμα των συστημάτων ασφάλισης που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική αρχή όσον αφορά τις αποζημιώσεις των επενδυτών. Εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι έτοιμες να αναλάβουν τέτοιες ευθύνες, τότε γιατί όχι. Εξάλλου, επιπλέον, είναι προφανές ότι η πλήρης κάλυψη των επενδυτών δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενό μηχανισμού που να βασίζεται στους κανόνες της αγοράς αποκλειστικά. Δεύτερον, για τα επίπεδα κάλυψης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ ότι οι πτωχεύσεις επενδυτικών οργανισμών, οι πρόσφατες, έδειξαν ότι τα επίπεδα κάλυψης λειτουργήσαν. Θέλουμε να αυξήσουμε το επίπεδο κάλυψης για τον κάθε επενδυτή. Είναι οι προτάσεις του Χόκμαρ και του Κεμάλ. Είναι ορθές και ανταποκρίνονται στην κατάσταση. Τρίτον, το επίπεδο εξάντε χρηματοδότησης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύω ότι είναι υπερβολική. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις προτάσεις της κυρίας Λούλινγκ. Νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να μιλάμε για ένα επίπεδο χρηματοδότησης εξάντε γύρω στο 0,1%. Αλλιώς τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα επίπεδα χρηματοδότησης ανάλογα με την πραγματικότητα που επικρατεί στην κάθε χώρα. Και όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο, νομίζω ότι είναι σημαντικό η περίοδος αυτή μεταβατική να είναι μεγαλύτερη. Η ιδεώδης κατάσταση θα ήταν ένα επίπεδο 10 ετών μεταβατική περίοδος. Όσο για το πεδίο εφαρμογή, συμφωνώ με την κυρία Μπέρες, μπορούμε να περιορίσουμε το επίπεδο προστασίας των επενδυτών στην αποζημίωση των σχετικών απολειών. για τα χρηματοδοτικά προϊόντα τα οποία εκδίδονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα ήθελα να επιμείνω ότι είμαι στη διάθεση όλων για συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κανένα άλλο ομιλητή δεν έχει ζητήσει το λόγο. Εκτό να επανέλθουμε στον εισηγητή, θέλετε να ακούσετε την άποψη τη Κομισιόν. Όλε. Πώς η Κομισιόν κάτι θέλει να πει, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε πέντε στοιχεία. Το πρώτο αφορά την εμβέλεια τη οδηγία. Κατά τη γνώμη μα, ε, θα πρέπει να υπάρχει πολύ ευρύ πεδίο για την οδηγία αυτή. Η Κομισιόν θα υποβάλει την πρόταση HOSITS 5, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γι' αυτό θα πρέπει να καθυστερήσει η συζήτηση τη αποζημίωση των επενδυτών, επειδή θα υποβληθούν νέε προτάσει που διακανονίζουν αυτό το θέμα το HOSITS 5, δεν θα υπάρχουν αργότερα. Όσον αφορά το θέμα της μείωσης του, του στόχου για την υποβολή εξάντα, ίσως χρειάζεται για να είναι λιγότερο ακριβό το σύστημα, να πρέπει να αλλάξουμε κάτι, αλλά εμείς προσπαθούμε να έχουμε μία δομή ουσιώδη. Η μείωση αυτή δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι υπερβολική. Όσον αφορά το σύστημα ασφάλισης, θα πρέπει να δούμε τελικά πώς θα λειτουργήσει το σύστημα της αποζημίωσης των επενδυτών. Το Φεβρουάριο οι υπηρεσίες Κομισιόν ε, προετοίμασε ένα μη έγγραφο, ένα non-paper που δόθηκε και στο Συμβούλιο και στον εισηγητή. Παίρνουμε ορισμένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείε για να αποφύγουμε να καταθούν πολύ ψηλά ποσά στα συστήματα τα οποία θα φερθούν από την οικονομία. Και θεωρούμε ότι θα υπάρχει κάποια δυνατότητα εισαγωγή κάποιων στοιχείων ασφαλιστικών αλλά πλήρη μεταφορά θα απαιτούσε περαιτέρω ανάλυση και όπως είπε και ο εισηγητής μια, ε, έναν έλεγχο των επιπτώσεων. Μετά, όπως ξέρετε, η μεταρρύθμιση του ΜΕΦΙΤ θα προταθεί από την Κομισιόν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. και εκεί ίσως θεωρήσουμε ορισμένοι από τους συγητές, από τους επενδυτές, συγγνώμη, που είναι επαγγελματίες επενδυτές, να χρειαστεί να αποσυρθούν από αυτό το κατάλογο. Η πρόταση που έχει υποβληθεί αυτή τη Κομισιόν προβλέπει ευθυγράμμιση ε, των σημείων για τους επαγγελματίες επενδυτές με το MIFID. Θα πρέπει λοιπόν να ασχίσουμε ε, τις προσπάθειές μας οριζόντια. Επίσης, ε, το θέμα της κάλυψης των ε, καταχρηστικών συμβουλών η πρόταση που υπέβαλε η Κομισιόν σχετικά επιτρέπει οι μηχανισμοί της αγοράς που υπάρχουν ήδη να παραμείνουν ε, επιτάπητος. Θα μπορούσε όμως να δημιουργηθεί ένα συμπληρωματικό κόστος, το οποίο δεν χρειάζεται σε κοινοτικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Όλε. Α, υπερβάσου. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Δηλαδή είναι πιο σημαντικό να έχουμε ένα μηχανισμό που να μην είναι ακριβώς, παρά να έχουμε μια καλή προστασία του καταναλωτή έναντι κακών συμβουλών, ανθρώπων που θα πουλήσουν σκάρτα προϊόντα. Τι λογική είναι αυτή. Εγώ δεν τη δέχομαι. Όλε. Όλες Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Υπάρχουν μερικά θέματα που πρέπει να τα δούμε και να βρούμε απαντήσεις ε, πιο σαφείς. Καταρχή δεν έχω αντίρρηση να μπουν και τα usage στην οδηγία αυτή. Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά τις πληροφορίες που έχω θα μου πείτε, μπορεί να μην, έχει σημασία για μερικούς από εσά. Καμία χώρα, ούτε μία χώρα δεν του ζήτησε αυτό. Και λένε να γίνει, να ρυθμιστεί αυτό στα usage. Το δικό μου το επιχείρημα, και για ποιο λόγο διστάζω να το δεχτώ αυτό που προτείνεται, είναι ότι θα στοιχήσει 27 δις ευρώ. Τεράστιο ποσό, κατά τη γνώμη μου. Και η Κομισιόν λέει ότι αυτό ε, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το κάνουν οι κακοί, όχι οι καλοί, λέει ο Σβέν. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, πες, πες ότι το είπα σαν αστείο. Ξέρω ότι ο ίδιος ο Επίτροπος και η Κομισιόν θέλουν να λυθεί το θέμα αυτό. Το συνάντησα και ξέρω. Και έχει τους λόγους του να το ζητάει αυτό. Και θέλει να συστρατευτούμε μαζί του. Αλλά η Κομισιόν, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να δώσει μερικές καλές απαντήσεις όσον αφορά το κόστος. γιατί το έχω ξαναπεί κάμποσες φορές στην Επιτροπή μας, δεν πάμε να εισάγουμε νέα νομοθεσία, νέες προτάσεις, χωρίς να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό στην αγορά. Και ο Επίτροπος μου λέει, εμένα, σε μένα, ότι προσπαθεί να κάνει μια μελέτη για τις 20 προτάσεις, πώς θα λειτουργήσουν, πώς θα επηρεάσουν την χρηματοδότηση. Στον κλάδο αυτό. Αν αυτό μπορεί να γίνει πριν ψηφίσουμε, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Το πρόγραμμα ασφάλισης. Είπα και πριν. Να το, να το δούμε. Αλλά κυρία συνάδελφε, θα πρέπει να δεχτείτε ότι έτσι ξαφνικά από μια στιγμή στην άλλη να πάρουμε ένα εντελώς νέο σύστημα και να πούμε αυτή είναι η σωστή λύση, αυτό δεν γίνεται. γιατί μας κατηγορούν ότι η νομοθεσία που βγαίνει από τα νομοθετικά όργανα δεν είναι απόλυτα κατανοητή. Γι' αυτό κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες για να δούμε αν και πώς θα λειτουργήσει αυτό. Οι κακή συμβουλή, κακές συμβουλές. Δεν έχω πιστεί Είχαμε προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι οι επενδυτές, εγώ ας πούμε, ως επενδυτής, έχουμε ευθύνη. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εισάγουμε αυτό το στοιχείο. Κύριε Μπερές, πιστεύετε ότι θα πρέπει να εισάγουμε το βρετανικό σύστημα στην Ευρώπη? Εγώ διστάζω. διάφορες οντότητες στις οποίες ε, αναφερθήκατε που προτείνατε από ό,τι ξέρω καλύπτονται από το MIFID. Αλλά να το δούμε. Ε, κάλυψα την ερώτηση του συναδέλφου Σάλμπα, της κυρίας Μπερές. Αν ήμουν διαιτητής που δεν είμαι, συνάδελφε, δεν θα είχατε κίτρινη κάρτα, θα έχετε κόκκινη κάρτα α, όταν είπατε για μένα ότι είμαι σοσιαλιστές. Δεν έχω τίποτα κατά των συναδέλφων που είναι σοσιαλιστές, αλλά είναι προσβολή για μένα. Και θα έπρεπε ενδεχομένω να αποφασίσει γι' αυτό η, η πρόεδρος. Α, ανέκδοτο ήταν γι' αυτό. Α, καλώς. Διαφάνεια. Καλό. Να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και νούμερα και αυτό καλό όπως είπατε. Χρήσιμο είναι για το πρόγραμμα ασφάλισης, απλώς χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Για τον Σβέν, για τα λόμπι, χρησιμοποιείς τον όρο αυτό. Είναι κακό? Όχι λες βέβαια. Γιατί χρησιμοποιεί την υποχιστόπιση. Λες και το λόμπι είναι κατά ανάγκη κακό. Εμένα κυβερνήσεις μου κάνουν λόμπι ένα ο κόσμος. Όπως είπε και ο κύριος Γκοζές, αν υπάρχουν καλές προτάσεις, γιατί δεν επιτρέπεται να τις εισάγουμε στο κείμενό μας. Να έχουμε μόνο μια δική μας, εντελώς δική μας εργαλειοθήκη, να είμαστε εμπειρογνώμονες επί των πάντων, δεν νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει καλύτερη νομοθεσία. Με τον κύριο Κλούτε. Συμφωνείτε. Ωραία. Χαίρομαι που συμφωνείτε. Κύριε Γκοζές, ήδη ανάφερα αυτό που είπατε και την κυρία Λούλινγκ. Είμαι υπέρ της πλήρους εναρμόνισης. Νομίζω αυτή είναι η τελικά η λύση. Ιδιαίτερα για αυτού του είδους προστασία του καταναλωτή. Ε, σημείωσα αυτά που είπε ο κύριος Φέιλ. Ευχαριστώ και την Κομισιόν με τις απαντη... για τις απαντήσεις της. Κλείνω με το εξής. Ήδη έχουμε μερικές συμβαστικές τροπολογίες. Θα σας μοιραστούν, θα τις μελετήσετε. Ο στόχος μου είναι να συμφωνήσετε όλοι, αν γίνεται. Αλλά για το usage και 150.000 είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε. Γιατί εγώ μένω, επιμένω στις 100.000. Δεν πρέπει να μειώσουμε την προστασία για ορισμένε χώρες. Αυτό είναι όμως και θέμα του Συμβουλίου. Και για τα usage είπα ήδη γι' αυτό. Αγαπητοί φίλοι, Σίγουρα στο τέλος θα έχουμε μια καλή πρόταση. Μισοφιλελεύθερη πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπως έχουμε ξεπεράσει τα χρονικά μας όρια, αλλά όλοι έπρεπε βέβαια να ε, ε, αμυθεί κατά όλων αυτών των κατηγοριών. Δεν ξέρω αν στο web stream θα καταλάβουν απαραίτητο τα ανέκδοτα και τα αστεία που λέμε εδώ συμφωνήσετε με το site για την πολιτική, αλλά όχι με την περιγραφή τη δική σας που έκανε από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων, η ψηφοφορία θα γίνει θεωρητικά στις 13 Απριλίου για να περνάσει στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Αυτό είναι ο στόχος και το μου τη της Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο τελικό θέμα τη μια για σήμερα. Η εξέταση της δέσμης για την οικονομική διακυβέρνηση. Ξέρω ότι οι συγητές ε, το συζητήσανε μεταξύ τους, αλλά αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε για να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Και ξέρω ότι όχι μόνο έχουμε καθυστέρηση, υπάρχουν και πολλά, πολλοί βουλευτές που έχουν υποβάλει τροπολογίες και θέλουν να μιλήσουν όπου θέλουν. Θα παρακαλώ στις ζητές λοιπόν να είναι κατά σύντομοι και να μην ξεπεράσουμε πέντε λεπτά ο καθένας. Εσείς Κορίν πρώτη. Thank you very much. And, uh, Ευχαριστώ πολύ. Και κόψτε με σε πέντε λεπτά. Ε. Έχω 559 τροπολογίες να εξετάσω από πολλούς συναδέρφους. Καταλαβαίνετε ότι θέλω να τους απαντήσω. Προηγουμένως όμως θέλω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ τη συνεργασία με όλους τους συναδέρφους. Είχαμε και πολύ καλή συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά και με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Να ξέρετε ότι κάθε φορά που έχετε μια ερώτηση για τις τροπολογίες σας, ελάτε να με βρείτε. Θέλω να είμαι ανοιχτή σε διάλογο μαζί σας, οπότε είμαι στη διάθεσή σας και εκτός αίθουσα συνεδριάσεων. είναι μια ισορροπημένη προσπάθεια που κάνουμε για να πετύχουμε μια ευρεία στήριξη του πακέτου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά εμένα, έχω την εντύπωση ότι θα πετύχουμε παρόλο που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα από ότι με το πακέτο εποπτείας, γιατί τα πράγματα τα οποία εξετάζουμε εδώ είναι θέμα έντονου ευρωπαϊκού συντονισμού, είναι θέμα του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επίσης υπάρχουν προκλήσεις ε, μεγάλες. Ε, έχουμε διαφορετικές πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαφορετικό υπόβαθρο κάθε φορά και διαφορετική οπτική γωνία ε, με την οποία βλέπουμε το πακέτο αυτό. Όσον αφορά τη δικιά μου την έκθεση, που είναι ε, επίσης μια πράξη ισορροπίας που προσπαθούμε να πετύχουμε, έχει πολλές τροπολογίες. Οι τροπολογίες αυτές τι ζητάνε. Ζητάνε μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά την εφαρμογή του 3% και του 60% κριτήριο χρέους και μιλάει για επενδυτικούς στόχους πέρα του 3%. Από την άλλη μεριά υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες περιορίζουν δεν αφήνουν καθόλου περιθώριο λιγμών μερικές φορές, ενώ υπάρχει κάπως την τρέχουσα πρόταση και ζητούν ε, περισσότερους κανόνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα νούμερα. Εγώ θα ήθελα να επιμείνουμε στην προϋπόθεση της φορολογικής σταθερότητας, γιατί αυτή είναι προϋπόθεση για ανάπτυξη. Οι διαφορετικές αλλαγές αλλάζουν την κατάσταση έχουν θετικές επιπτώσεις. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση μας βρίσκουν βέβαια σύμφωνους. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ε, ε, προληπτικής ε, πολιτικής, εγώ προσωπικά έχω μία διατύπωση η οποία αναφέρεται στην διόρθωση μέσοπρόθεσμα, βάσει δηλαδή των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων. Ασχοληθήκαμε επίσης και με διάφορες τροπολογίες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τον κυκλικό χαρακτήρα. Όσον αφορά τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, θέλω να αναφερθώ στις τροπολογίες του Οτομπούμαν Μπούμαν και αλλωνών που μιλούν για επενδυτικούς στόχους. Εδώ έχουμε μια δυσκολία. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω αυτή την τροπολογία και είναι σαν να ξαναμπαίνει ο, κανόνα, ο χρυσός κανόνας. Ήταν κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει και στα πλαίσια της συνθήκης του Μάστριχτ τότε. Τότε είχε απορριφθεί, γιατί σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν επιπλέον επενδυτικούς στόχους πέρα του 3% δηλαδή. Αν το κάνουμε αυτό, τότε ε, διακινδυνεύουμε την εμπιστοσύνη στο πακέτο ολόκληρο. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τρισέ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χτες ήταν ξεκάθαρος. Είπε ότι είναι επικίνδυνο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να καθίσω και να σκεφτώ με τους συναδέρφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες για να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε πιο μεγάλη δέσμευση προκειμένου να πετύχει η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Ναι, αλλά να μην δούμε μόνο τις επενδύσεις, να δούμε και την κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση της απασχόλησης στα κράτη-μέλη επίσης. Και αυτά πρέπει να τα δούμε. Ήδη στην οδηγία υπάρχει ένας προσωρινός αποκλεισμός Υπάρχει ήδη στην οδηγία μια απόκληση, συγγνώμη, γι' αυτό. Και θα ήθελα αυτό να το διευκρινίζουμε περισσότερο. Επιπλέον, να έχουν ήδη περάσει τα πέντε λεφτά. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο τώρα και τα εθνικά σχέδια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι πιο έντονο στην πρόταση γιατί τότε πετυχαίνουμε μια πιο ολοκληρωμένη κάλυψη. Θα ήθελα να μιλήσω και για την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία. Υπάρχουν τροπολογίες που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να τονιστεί το θέμα των ε, δαπανών. Ε, γι' αυτό το εγώ το βάζω επίσης, αλλά κάπως πιο ήπια το διατυπώνω. Δεν μιλάω για περικοπές. Λυπάμαι που δεν έχω περισσότερο χρόνο, θα ήθελα να σας εξηγήσω και άλλα πράγματα. Ίσως στο τέλος άμα μείνει χρόνος, λέει η Πρόεδρος, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι κι αλλιώς τον χρόνο που έχουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Περνάω στον Διέγκο τώρα. Σε σχέση με, με, το, με τη δική μου έκθεση, σχετικά με τις διορθωτικές διαδικασίες μέσα στα πλαίσια του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας υποβλήθηκαν πάνω από 300 τροπολογίες όσον αφορά τα άρθρα είναι δυνατόν σε μια πρώτη φάση να κάνουμε μερικές ε, συμβαστικές ε, προτάσεις, πάνω από 15. Πιστεύω ότι οι ιδεολογίες, οι τροπολογίες για τις αιτιολογικές σκέψεις θα είναι κάπως πιο εύκολο. Εφιστώ την προσοχή σας στα εξή πέντε σημεία που είναι τα πιο δύσκολα, τα πιο λεπτά σημεία. Το ένα αφορά τον ρυθμό μείωσης του ελλείμματος. και το ποσό της μείωσης. Γιατί έχουμε πολλές διαφορετικές προτάσεις. Μερικοί συνάδελφοι από την ομάδα των φιλελευθέρων θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει μείωση στο 1 εικοστό αλλά στο 1 δέκατο. Και θεωρούν ότι αυτή η μείωση πρέπει να γίνει σε δύο χρόνια και όχι σε τρία. Άλλοι συνάδελφοι από τη σοσιαλιστική ομάδα θεωρούν ότι αυτή η μείωση πρέπει να είναι στο 20 για περίοδο τριών ετών με δυνατότητα να υπάρχουν και εξαιρέσει όταν το νέο χρέος οφείλεται σε δημόσιες επενδύσεις. Άλλοι θέλουν να το συσχετίσουν με άλλες παραμέτρους. Εγώ προτείνω το εξής. Μέσο όρο τρία χρόνια για τη μείωση του ελλείμματος γιατί το θέμα είναι πολύ επίδικο και θα προσπαθήσω να πετύχω ένα συμβασμό μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντως θα ισχύσει αυτό που ισχύει στο Κοινοβούλιο, δηλαδή ο δημοκρατικός κανόνας στην ψηφοφορία. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα των ποσοστών. Σε σχέση με τις εξαιρέσεις. Και εδώ έχουμε πολλές διαφορετικές προτάσεις. Είτε προτάσεις που κινούνται προς τα κάτω, χαμηλά, 0,03% του ΑΕΠ και προτάσεις οι οποίες είναι πιο μαξιμαλιστικές όπου οι εξαιρέσει καλούνται να είναι το 0,4% με μέγιστο 1% του ΑΕΠ. Τρίτο θέμα το ετήσιο ποσό μείωσης του ελλείμματος. Όταν έχει κινηθεί η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η Κομισιόν έχει κάνει μία πρόταση με ελάχιστο ποσό 0,5%. 0,5. Υπάρχουν συνάδελφοι που έκαναν εναλλακτικέ προτάσεις, μείωση 1% ή μινιμαλιστικές προτάσεις, μείωση 0,2%. Σας θυμίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι ιδιαίτερα ακαθόδης διότι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ε, τα επιχειρήματα που βρίσκονται πίσω από την κάθε μία πρόταση. Μερικές φορές προτάσεις αυτές είναι αυθαίρετες, άρα είναι δύσκολο να πετύχουμε συμβιβασμό. Τέταρτο μεγάλο θέμα, η κατακαιρματισμένες προτάσεις. Τι εννοώ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλους τους παράγοντες που θα πρέπει να μπουν στην ε, έκθεση για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Και τέλος, πέμπτο, οι εξαιρέσει λόγω δημοσίων επενδύσεων και ποιας ποιότητας πρέπει να είναι αυτές οι επενδύσεις. Αυτά είναι τα πέντε μεγάλα θέματα. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο τελικά θα συμφωνήσει σχετικά με την κοινοτική μέθοδο και δύο παρατηρήσεις για να τελειώνουμε αυτή την εισαγωγή. Η συζήτηση με τους άλλους σκιώδεις συγητές μέχρι στιγμής πήγε καλά. Η δυνατότητα να μπει η διαδικασία αυτή στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 στο Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, σας θυμίζω ότι αυτό αποτελεί για μας μεγάλη πρόκληση. Μένουμε λοιπόν με τις προτάσεις του Σεπτεμβρίου ή αν θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι ας βάλουμε στο πακέτο αυτό πολλά από αυτά τα στοιχεία που τα συζητάνε ήδη οι πολίτες μας συνεχώς. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η Ελίσσα έχει το λόγο. Θα μιλήσω, θα μιλήσω αγγλικά. Και εγώ θα αναφερθώ σε πέντε θέματα για το μακροοικονομικές ε, ανισομέρειες. Το πρώτο είναι η ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε ανισομέρειες. Οι συνάδελφοι που έχουν κάνει προτάσεις νομίζω έχουν δίκιο. Πιστεύω ότι θα βρεθεί συμβασμό. Το δεύτερο, οι μακροοικονομικές ανισομέρειε και οι δείκτε οι ίδιοι. Μερικοί συνάδελφοι ζητάνε να μην μπει τίποτα το κοινοβούλιο γι' αυτό. Βλέπουμε όμως ότι σιγά σιγά ορισμένες παράμετροι που θα έπρεπε να μπουν σε αυτό εδώ το βαθμολόγιο scoreboard να τα συζητάνε διακυβερνητικά. Και πέρασαν σε αυτό που το λέμε σύμφωνα για το ευρώ ή σύμφωνα για Το να θέλουμε οι παράμετροι αυτοί να μπουν υπό την κοινωτική μέθοδο και νομική βάση συζητιόνται όλο και περισσότερο τώρα ο κύριος Τρισέ ή Κομισιόν μας λένε ότι αυτό έχει νόημα. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει ομοφωνία εισάγοντας μερικά από τα στοιχεία που αυξάνουν την κατανόηση της κατάστασης στις διάφορες χώρες. Τρίτο σημείο. Το σύνολο δικτών. Θα πρέπει να φροντίσουμε να επιτευχθεί σωστή ισορροπία. Μεταξύ των συναδέλφων που πρότεινα να μπουν πάρα πολλοί δείκτες που να καλύπτουν πάρα πολλά θέματα και από την άλλη μεριά να έχουμε δείκτες, η θεωρία που λέει να έχουμε δείκτες που είναι διαχειρίσιμοι μέχρι 12 το πολύ Οπότε να ξεφύγουμε από τα θέματα βραχυπρόθεσμης σύγκλησης. Ελπίζω να πετύχουμε συμβασμούς με τους σωστούς δείκτες με ευελιξία, με καθολικότητα, με ευρύτητα, να καλύπτει η πραγματική οικονομία, η απασχόληση, η ανταγωνιστικότητα. και με καλύτερη κατανόηση της κατάστασης της κάθε μιας χώρας. Τέταρτη ομάδα θυμάτων είναι ο ρόλος του βαθμολογίου, του συγκριτικού βαθμολογίου scoreboard. Μία σειρά δικτών για ανάλυση από την Κομισιόν και από την Κεντρική Τράπεζα όπου θα πάνε και θα συζητάνε στην κάθε μία χώρα τις συστάσεις τους και το πακέτο αλλαγών που θα πρέπει να εισάγει η χώρα. Όχι με αυτόματο χαρακτήρα, όχι με προκαθορισμένες συνταγές. Αυτό συμφωνεί με την περιγραφή που μας έκανε η Κομισιόν το πρωί σε μια σημαντική συνάντηση όπου ο Επίτροπος μας περιέγραψε αυτό το νέο σετ δικτών τις μακροοικονομικές ανισορροπίες ως ένα καλό σετ για ανάλυση δύσκολο μεν αλλά πιο γόνιμο. Εδώ τίθεται και θέμα συμμετρίας. Βέβαια διαφορετική ερμηνεία θα έχουμε αν έχουμε πλεόνασμα ή αν έχουμε έγκλημα. Και τέλος, επειδή όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε και να κάνουμε συστάσεις, Γι' αυτό εγώ λέω όχι αυστηρές κυρώσεις. Μια συμβολική ποινή είναι υπέρ της θέσης της Κομισιόν. Εγώ και ο Καρλ Άγγλουντ έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ στενά και, θεωρώ ότι σε μια δύσκολη στιγμή όπως αυτή εδώ και ένα δύσκολο θέμα όπου και η Κομισιόν έχει δυσκολία να κάνει έντονες συστάσεις για την αγορά εργασίας, για την έρευνα και την ανάπτυξη, για τη χρηματοδότηση. Πρέπει να προσέξουμε να μην ξεπεράσουν τα λογικά όρια προκειμένου να επιτευχθεί ένας αυτοματισμός. Δηλαδή, να δώσουμε στο σύστημα χρόνο να λειτουργήσει, προσεκτική με το μηχανισμό κυρώσεων. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έστειλαν υλικό στην έκθεση. προσπαθώ να πετύχω σωστές και καλές συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη Σιλβή. Ευχαριστώ Σάρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και εγώ έχω 250 τροπολογίε για το κείμενο αυτό, τεράστια συλλογική εργασία. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε ε, μετακινείται συνεχώ ε, δεδομένων των συναντήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ευρωζώνη, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για του 27 κλπ. Στα σύντομα. Εγώ έχω ένα κείμενο που αφορά το ποινικό δίκαιο, κύριο κλπ. Όσον αφορά αυτή την πτυχή του ποινικού δικαίου, ομολογώ ότι η κοινωτική μέθοδος είναι καλή και η Κομισιόν προτείνει κάτι που είναι σχετικά ισορροπημένο και οι τροπολογίες ε, είτε πιο μαξιμαλιστικές είτε υπερβολικού περιορισμού ε, μπορούμε να σκάνουμε να παραμείνουμε ευθυγραμμισμένοι με αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Κατεβλήθησαν προσπάθειες ε, δημιουργικότητας. Ευχαριστώ τον Φιλίπ Πλομβέρ ιδιαίτερα που προσπάθησε να προτείνει κάτι που θα ήταν ε, σαν μια άδεια με πόντους ας πούμε που τη βρίσκω πολύ ελκυστική. Απ' την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι όλοι οι συγκητέ πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Δηλαδή, προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι πριν από το καλοκαίρι, όπω μα το ζητάει το Συμβούλιο, δεδομένου ότι υπάρχει μια δέσμη σαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και είναι δύσκολο να το εφαρμόσουμε αυτό. Απ' την άλλη μεριά θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιό κατά πόσον πραγματικά ε, επιμένει σε αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ ικανοποιητικό σύστημα κυρώσεων μακροπρόθεσμα. Δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι η εργασία της Κορίνη για την πρόληψη, η εργασία της ε, Ελίζα θα μας ε, κάνει να αποτρέψουμε τις κυρώσεις. Αν φτάσουμε στις κυρώσεις όμως έχουμε ένα ε, σύστημα το οποίο είναι πολύ ελάχιστο. Επίσης δεν έχω ακόμα κυκλοφορήσει τον απολογίες συμβασικές, γιατί είχαμε σημερινή όπου αναπτύχθηκαν ε, τα, το θέμα των ευρωομόλογων ε, την περασμένη εβδομάδα και ευχαριστώ στους συναδέλφους που ήταν παρόντες. Ε, η οικονομολόγη αυτή και ευχαριστώ και τη γραμματεία για την εργασία των πυρογνωμόνων για το θέμα αυτό. Υπάρχει, λέω, μια σχετική σύγκληση όσον αφορά το χρήσιμο οικονομικά χαρακτήρα για το ευρώ, να δημιουργηθούν δηλαδή κάποια μέσα που δεν σέβονται το, την πειθαρχία και υπάρχει και μία ομοφωνία όμως όσον αφορά τα νομικά εμπόδια, κλασικό δίλημα δηλαδή, του ευκταίου και του δυνατού. Και ξέρω ότι πολλοί ε, συνάδελφοι από βόρειες χώρες μου είπαν ότι γίνεται στη Βλανδία, στη Γερμανία κλπ. Έχω πολύ σεβασμό για τη δύσκολη πολιτική συζήτηση στο ιστορικό των χώρων αυτών. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή ΕΚΟΝ να παραμείνουν προσκολλημένοι στην ε, υποβληθήσα πρόταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καθένας από εμά να συμπεριφερθεί σαν βουλευτής του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ακούσει δηλαδή τους εκλογές του, αλλά να καταλανοήσει και τους περιορισμούς που έχουν άλλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, μειώσουμε αυτή την αντιπαράθεση βορρανότου που είναι πολύ δυσάρεστη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν αρνούμεθα, και το είπα χθε τον κύριο Τρισέ, δεν αρνούμεθα κάποια πράγματα επειδή μας λένε δεν είναι δυνατό. Αν το είχαμε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε το ευρώ. Γιατί ε, αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα αν είχαν ακολουθηθεί οι πεσημιστές τότε. Προσπαθώ να ακολουθήσω πολλές από τις προτάσεις. Στη χώρα μου πολλοί δεν συμφωνούν, αλλά πρέπει να έχουμε κάποια μεσοπρόθεσμα στοιχεία στη δέσμη πέρα από αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε θα συμβάλλουμε στην συλλογική εργασία και ευχαριστώ για άλλη μια φορά την Γραμματεία και του συναδέλφου γιατί εργαζόμαστε με πολύ καλή ατμόσφαιρα παρόλο που τα θέματα αντικειμενικά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σε ευχαριστώ και ούτε καν αυτά τα πέντε λεπτά. Θαυμάσιο. Ο Καρλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να μην φτάσω στα πέντε λεπτά. 200 τροπολογίες είχα που με ικανοποίησαν που οι περισσότερες για να είναι πάρα πολύ επικοδομητικές και προσβλέπω πραγματικά να ενισχύσουν όλα τα τμήματα της ε, ε, μακροοικονομικής εποπτείας. Καταρχήν το θέμα που θα ήθελα να εξετάσω είναι η, τα πρόστιμα το επίπεδο των προστήμων και πώς θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε πάνω σε αυτά. Αυτό είναι κάτι που απασχόλησε πολλούς και οδήγησε στις εξελίξεις που είναι κατανοητές ίσως. Και υπάρχει ε, αυτό το, αυτή η διαπραγμάτευση όλων λέει 0,4, άλλος λέει 0,2, άλλος λέει κατά διάμεση στα 2 και θα πρέπει να αναλύσουμε να δούμε ποια είναι η πιο σοφή μέθοδος. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε μια λύση. Υπάρχει ευρία κατανόηση νομίζω στο θέμα αυτό. Μετά υπάρχει και όλη η διαδικασία λήψεων αποφάσεων όσον αφορά τα πρόστιμα και την επιβολή τους. Σε πολλούς τομείς αναφέρεται η ψηφοφορία με σταθμισμένη πλειοψηφία, αλλά είναι καμιά φορά προβληματική. Και υπάρχουν και συνάδελφοι που προτείνουν η Κομισιόν να πάρει αυτές τις αποφάσεις για την υποβολή και να μην εμπλεκεί καθόλου το Συμβούλιο. Ενδιαφέρουσα σκέψη, σκληρή όμως. Κάτι άλλο είναι το τι θα γίνει με τα χρήματα αυτά που συλλέγονται ενδεχομένω από πρόστιμα. Ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί, αλλά εάν, πού θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Και τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία συνένεση τα χρήματα αυτά να δοθούν στη ΕΦΣΕΦ και αργότερα στο μόνιμο σύμφωνο σταθερότητας η πράσινη συζήτηση ότι θα πρέπει να το βάλουν τα χρήματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν είναι δυνατό. Πρέπει βέβαια να δούμε τι γίνεται με αυτό το νέο μηχανισμό που πρόσφατα, χθε δηλαδή, ε, συστήθηκε αναλυτικά στην, στο Συμβουλίο Κοφίν. Ένα άλλο θέμα είναι τα πρόστιμα για την χειραγώγηση στοιχείων. Υπάρχει νομίζω ευρεία συμφωνία ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις για χώρες οι οποίες δεν δίνουν επαρκή και σωστά στοιχεία. Βέβαια το θέμα είναι ότι πώς θα ορίσουμε ότι κάποιοι έχουν χειραγωγήσει αυτά τα στοιχεία. Ε, υπάρχει και κάποια πρόκληση. Άλλα θέματα που ίσως αξίζει να αναφερθούν αυτή τη στιγμή είναι το ότι είναι οι εξαιρετικές οικονομικές ε, προϋποθέσεις. Το θέμα της εθνικής ιδιοκτησίας, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους για όλες εκθέσεις. να δούμε πού είναι χρήσιμο και κατάλληλο να εμπλακεί το κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή. Και για λόγους διαφάνειας, αλλά και για λόγους λήψης απόφασης. Έχουμε τον σημαντικό ρόλο λοιπόν να παίξουμε. Και τέλος, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι εργαζόμαστε με συνέπεια. Γιατί πολλά από τα τμήματα του δικού μου κειμένου εξαρτώνται από κάποια τμήματα στα άλλα κείμενα. Πρέπει να είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι. Τούτων εκθένων είμαι πολύ ευτυχής για την πολύ επικοδομητική ατμόσφαιρα συνεργασίας που είχαμε. Αυτά με δύο λόγια. Και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ευρεία συνένωση. Τέλος, ορισμένοι έχουν προτείνει να διαγραφεί όλη αυτή η νομοθεσία. Δεν ξέρω ε, Κατά πόσο μπορούμε το έχουμε συμβασμού, αλλά αυτή είναι η τελική γραμμή. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κάρλ. Η Βίκη, τέλο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους συναδέρφους που κράτησαν τις τροπολογίες τους κάτω από 200. Οι τροπολογίες όλες ήταν πολύ <clears throat> ενδιαφέρουσες, Έχω κάποιες συμβαστικές να προτείνω, δεν ξέρω αν τις έχουν δει όλοι. Βασίζομαι πρώτα απ' όλα στα, στις λογιστικές προδιαγραφές και στην ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες προδιαγραφές, ε, ρευστού και όχι. Έχουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλάει για στοιχεία με νούμερα. Μιλάει για τις τοπικές κυβερνήσεις. Δεν ξέρω η Άστριτ. Α, Άστριτ. Άστριτ. Άστριτ, μ' ακούς? Κυρία Λούλινγκ. Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε η 125 τροπολογία σας ε, τι ακριβώς εννοεί. Όσον αφορά τώρα τις προγνώσεις, ποιος είναι υπεύθυνο για τις προγνώσεις. και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στα κράτη, στις προγνώσεις των κρατών μελών και στις προγνώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή προφανώς προσπαθεί να συγκεντρώσει προγνώσεις που να έχουν κάποιο νόημα μεταξύ 27 χωρών. Δύσκολο. Εγώ προτείνω ένα συμβιβασμό που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον το επιθυμούν, να μπορούν να το κάνουν. Πολύ βασικός είναι ο έλεγχος για την πρόγνωση και το λέμε και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για την Ευρωζώνη. Πολλές τροπολογίες είχα επίσης που ζητούν ένα ανεξάρτητο σώμα να αναλαμβάνει ρόλο και στην ε, πρόγνωση και στην εφαρμογή των φορολογικών κανόνων. Τώρα η διατύπωση για τα ανεξάρτητα ε, για τους ανεξάρτητους αυτούς ε, οργανισμούς έχει βγει από το κείμενο του Συμβουλίου παρόλο που εμείς το θέλαμε υποχρεωτικά για την Ευρωζώνη. Φαντάζομαι ότι θα βρούμε κάποιο συμβιβασμό. Ίσως αν υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα στην Ευρωζώνη. Συνένεση τώρα για τους ε, κανόνες με την αριθμητική έκφραση, τους ταμιακούς. Και εδώ υπήρχαν πολλά σχόλια. Γενικά μιλώντας πάντως υπάρχει συνένεση ώστε να έχουμε μία οδηγία που να μπορεί να λειτουργήσει, να λαμβάνει υπόψη το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τις πληροφορίες που έρχονται ως πρόγνωση με μια μεθοδολογία που να είναι αξιόπιστη και να βασίζεται σε ανεξάρτητες εκτιμήσεις γιατί αλλιώς δεν θα καθυσυχαστούμε. Η βασική αρχή είναι να έχουμε τέτοιες καλές προγνώσεις που να μην χρειάζεται να ανησυχούμε από εδώ και πέρα. Πάντως, εδώ πέρα το κεντρικό σημείο δεν είναι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Πάρα πολλές τροπολογίες προσπαθούν να επαναλάβουν ε, την συζήτηση για το άγγραφο της Κορίν, την έκθεση της Κορίν ποιότητα δημοσίων δαπανών, πρόστιμα για τα κράτη-μέλη. Όχι, δεν έχουν θέση σε αυτήν την οδηγία. Σε κάποιο άλλο σημείο. Πρόκειται για πακέτο έξι εκθέσεων. Εδώ πρέπει να περιοριστούμε στα θέματα που θέλουμε να καλύψουμε και όχι να μπούμε σε κάτι γενικότερο, κατά πόσο οι δημόσιες δαπάνες γίνονται καλά ή δεν γίνονται καλά κλπ. κλπ. Να μην μπουν αυτά τα πράγματα σε αυτή την οδηγία. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως όλους και τον όγκρο συνάδελφο για τροπολογία 135 ήθελα κάτι να ρωτήσω, αλλά δεν βλέπω να είναι εδώ. Έχω μακρύ κατάλογο μιλητών, λέει η πρόεδρος. Θα σας πω, η κυρία Χιούμπνερ έτσι κι αλλιώς πρέπει να φύγει και είναι σκιώδης, οπότε, Ντανιούτα, για ξεκίνα εσύ και μετά θα πω ποιοι είναι στο κατάλογο μιλητών. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Χούμπνερ, για το βαθμολόγιο. Είναι το ένα που θέλω να πω και το άλλο έχει να κάνει με τις κυρώσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι αν δει κανεί τι τροπολογίε, υπάρχουν διάφορε επιλογέ για το βαθμολόγιο. Είτε ένα κατάλογο δικτών, πολύ μακρύ όμω, ή μπορούμε να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει για ένα σύνολο δικτών ε, βάσει πράξεων κατεξουσιοδότηση. Αν προτιμήσουμε τις ή πράξεις, τότε οι δείκτες πρέπει να μείνουν στη διαδικασία αυτή και όχι στον ίδιο τον κανονισμό. Καλό θα ήταν να μην είχαμε και τα δύο, και η πράξη, αλλά και έναν μακρύ κατάλογο δικτών στον κανονισμό. Ο κατάλογος δικτών που έχει ήδη μέσω τροπολογιών είναι λόγος ανησυχίας κατά τη γνώμη μου. Γιατί αυτά που προτείνονται αποτελούν μέρος ε, στόχων γενικότερης οικονομικής πολιτικής και καλύπτονται από το άρθρο 121. Η επιλογή των δικτών που θέλουμε εμείς πρέπει να έχει να κάνει μόνο για την εποπτεία εσωτερικών και εξωτερικών ανισορροπιών, προβλήματα ανταγωνισμού, υπερβολικό δημόσιο χρέος κτλ. Θα έπρεπε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις ή πράξεις και όχι τον κανονισμό. Έρχομαι τώρα στα μέτρα συμμόρφωσης για να διορθωθούν οι ανισορροπίες. Έρχονται στο παιχνίδι όταν έχουν χάσει τα κρατη δύο προθεσμίες ήδη και δεν προβλέπεται τίποτα, κανένα μέσο για τις χώρες εκείνες που έχουν χάσει την πρώτη προθεσμία να μπορεί να γίνει κάτι. Και τώρα έχει χαθεί και η δεύτερη. Άρα τι νόημα έχει να βάζουμε χρονικά όρια και προθεσμίες. Γι' αυτό και προτείνω τροπολογίες έτσι ώστε να προβλέπετε κάτι για τις χώρες εκείνες οι οποίες ε, δεν τηρούν τις προθεσμίες. Και μετά την ε, δεύτερη παράβαση της προθεσμίας, τότε εφαρμόζονται πρόστιμα. Έτσι νομίζω ότι θα ήμασταν πιο αποτελεσματικοί στη διαδικασία. Η πρώτη προθεσμία έχει ένα πειθαρχικό ρόλο. Τα κράτη-μέλη μπορεί να αποφασίσουν μετά την πρώτη προθεσμία να αποφύγουν τη δεύτερη. Αλλά αν φτάσουμε στη δεύτερη παράβαση είναι πολύ πιο εύκολο να πεις ότι βάζεις πρόστιμο στις χώρες αυτές. Έτσι νομίζω ότι είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πριν πω ποιοι είναι οι ομιλητές, θέλω να σας πω ότι ΑΦΚΟ ομόφωνα ενέκρινε ένα συμβαστικό κείμενο μετά τις διαπραγματεύσεις που είχε με το Συμβούλιο και με τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για τις αλλαγές στη συνθήκη. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 3. Τέταρτη, ναι. Τετάρτη, ναι. Ε, δεν κάνω εγώ λάθος, όντως Στι 3 εκτάκτος θα γίνει η ψηφοφορία αυτή αύριο στην Ολομέλεια. Δεν θα μπω στι λεπτομέρειε, πάντως αποφάσισαν πάνω στο τελικό κείμενο, δεν υπάρχουν τροπολογίε, έτσι κι αλλιώ η προθεσμία ήταν χτε. Έρχομαι στο κατάλογο μιλητών. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να μιλήσουν. Θα προσπαθήσω να έχω πρώτα τους σκιώδεις, που σημαίνει ότι ορισμένοι που νωρί ζήτησαν το λόγο, όπως η Περβάν και ο Γκουγκούνερ, θα πάρουν το λόγο αργότερα γιατί δεν είναι στοιχειώδης. Έχω. Philip Lamberts, Mr. Karins, Liam Wangok, Jürgen Klut, Edward Cicluna. Edward, you... Edward, και εσύ. Dorfman, then, then Gunnar and Pavanch and Ola Ludvigsen. So anybody else? Άλλος κανείς. Α, μετά. Α, η Άστριντ. Έχω ένα ραντεβού στις 6. Και έχω ζητήσει το λόγο. Θα δώσω αυτό που θέλω να πω γραπτά στην Βίκη Φόρτ. Καλώς, λέει πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ούντο. Ευχαριστώ, ε, αναφερθούμε δύο-τρεις φορές στο πολιτικό αποτέλεσμα που πρέπει να πετύχουμε. Ε, εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Τρουσέ για τις δυνατότητες των αντιμετώπισης κρίσης, αλλά όταν εμείς στην Επιτροπή έπρεπε να του επιβάλλουμε τι θα πρέπει να κάνει στο μέλλον όσον αφορά την ε, πολιτική επιτοχή ή τι θα πρέπει να κάνει στο μέλλον ε, υπέρ κατά, θα έλεγε αυτό είναι δική του ευθύνη. Και ακριβώς το αντίθετα αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορεί να βγει κανένα από τη διαδικασία αυτή και την επόμενη φορά να σταθεί ενώπιον των εκλογών στι ευρωεκλογέ και να πει ότι το αποτέλεσμα τη μεταρρυθμίση του Συμφώνου ε, Σταθερότητας και ανάπτυξη είναι ότι ακολουθήσαμε τον κύριο Τρεσέ. Όχι. Η κύριε Φέο, η κυρία Βόλμαν ε, ε Κολ, κύριε Κουλάρ θα πρέπει να ε, πείσουν τους εκλογείς ότι ήταν λογικό αυτό που κάναμε και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Κατόπιν, ε, όταν αναλύουμε γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι κυρίως, δεν είναι κυρίως ή αποκλειστικά, τονίζω, η ευθύνη στα κράτη-μέλη που, κάνουν, ε, που χρεώνονται ανεύθυνα. Όχι. Κατά βάση είναι πάρα πολύ κακοί κανόνες για την, ε, το τραπεζικό τομέα, οι ανισορροπίες που μόνιμα υπάρχουν στην Ευρωζώνη από την οικονομική κατάσταση και η αδυναμία η κοινωνία να ξεχρονιστεί πολιτικά και κοινωνικά. Και θα πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούμε ε, συνετά και εφιώς. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ δεσμευμένοι σε μια πολιτική παγίωση. αλλά εκτός από μια πολιτική κυρώσεων έχουμε και μια πολιτική με κίνητρα. Θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη να πραγματοποιήσουν καλές επενδύσεις, να αναλάβουν τις προσπάθειες εξυγχρονισμού που χρειάζονται, που είναι η παιδεία, αλλά όχι μόνο, είναι και ενέργεια και άλλα. Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μετά την Ιαπωνία θα έχουμε μια τελείως διαφορετική συζήτηση για την ενεργειακή πολιτική από την πριν από την Ιαπωνία, αλλά θα απαιτήσει αυτό μεγάλες προσπάθειες και δεν πρέπει να προσποιούμε ότι δεν είναι επιτάπητο στο θέμα. Θα πρέπει να δούμε να υπάρχει ε, μια αξιολόγηση καλών επενδύσεων του 2020 γιατί το σύμφωνο δεν επιτρέπεται να μην τα αναγνωρίζει, δεν επιτρέπεται να τις βάζει επίσης όρις όπως ε, ε, πολιτικές ε, παράλογες δαπάνες και θα πρέπει να εξετάσουμε λογικά σε ποιο σημείο του κύκλου της οικονομίας ε, βρισκόμαστε. Κακή πολιτική δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Ε, αν τα πετύχουμε όλα αυτά που τα επιδιώκουμε με τις δικές μας τροπολογίες, θα πετύχουμε έναν καλό συμβασμό στον οποίο είμαστε διαθέσιμοι να συνεργαστούμε. Αυτό που δεν θα κάνουμε είναι ότι δεν θα είμαστε στη διάθεσή σας για έναν κακό συμβιβασμό που δεν μπορούμε να προασπίσουμε ενώπιον των εκλογέων. Και γι' αυτό συζητάμε μαζί σας συνάδελφοι για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ Φιλίπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο σύντομε παρατηρήσεις Πρώτα για τη Σιλβή. Ω συμπρόεδρο των Πρασίνων, Ευρωπαίων Πρασίνων, και εγώ θεωρώ εκπροσωπώ ότι όλου του Ευρωπαίου πολίτε και μόνο των χωρών μα, τη χώρα μου. Γι' αυτό με ενδιαφέρει και η γνώμη του Γερμανού φορολογούμενου και η γνώμη του νεαργού Ισπανού άνεργου. Όλοι οι πολίτες το αξίζουν αυτό. Δεύτερον, ως ε, Ευρωπαίος Φεντεραγιστής, επαναλαμβάνω ότι ναι μεν να δώσουμε περισσότερες εξουσίες στην Κομισιόν σε ένα ουδέτερο όργανο, άξιο εμπιστοσύνη η συμπεριφορά της Κομισιόν, ιδιαίτερα με βάση την ετήσια έκθεσή της, κάνει ζημιά στην εμπιστοσύνη που της έχουμε. Γιατί η έκθεση αυτή είναι πολύ ιδεολογικά χρωματισμένη που ρίχνει το μεγαλύτερο βάρος στην προσαρμογή εντός εισαγωγικών που πρέπει να την πληρώσουν οι μέσοι πολίτες και εργαζόμενοι. Ε, μια πρώτη προσπάθεια με συμβαστικές τροπολογίες. Δεν θα διαπραγματευτώ εδώ το θέμα αυτό, απλώς θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Πρώτον, σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε ισορροπία στους προπολογισμού, όχι μόνο τις δαπάνες. Κάθε φορά που μιλάμε για δαπάνες θα πρέπει να συμπληρώνονται, να αντισταθμίζονται με τα έσοδα. Και όταν δεν μιλάμε για έσοδα, τότε να μην μιλάμε και για δαπάνες. Να μιλάμε μόνο για ισοζύγιο. Δεύτερον, η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια ανάλυση για ελαφρυντικά. Μερικοί θέλετε το σύμφωνο αυτό να λειτουργεί με αυτοματισμό. Εμείς θέλουμε να λαμβάνει υπόψη, να λαμβάνει υπόψη όλος ο επιχειρηματικός κύκλος. Μερικοί από εσά μιλάτε για μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και άλλα πράγματα, παραδείγματος επενδύσεις που θα μειώσουν το βάρος που θα φέρουν μελλοντικέ γενιές. Το επόμενο το σύμφωνο σταθερότητας ανάπτυξης. Ο κανόνας του ενός εικοστού, η μείωση του χρέους, ίσως να είναι ο παράγοντας ο οποίος να συντρίψει όλους τους άλλους. Δέστε μερικές χώρες μέλη τι συμβαίνει. Αυτός είναι ο κανόνας ο οποίος θα συντρίψει χώρες και πολιτικές και δεν θα βγούμε από την κρίση ποτέ. Αν δεν υπάρχει ρεαλισμός στην εφαρμογή αυτών των κανόνων θα είναι πολύ δύσκολο για μας να δεχτούμε αυτό το πακέτο. Τέταρτο, οι μακροοικονομικές ανισομέρειες. Μερικές χώρες μας ζουν μια κατάσταση που την ξέρουμε. Δέστε τι γίνεται με την Ιαπωνία. Όλοι αντιδρούν, λες και η Ελλάδα είναι το παράδειγμα, η κακή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και όλοι οι άλλοι είναι αθώοι. Δεν συμβαίνει αυτό. Ο πολίτης στην Ισπανία και την Ιρλανδία είναι, δεν είναι η μόνη ένοχη. Και σε δικές σας χώρες και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συμπεριφέρθηκαν τελείως ανεύθυνα και πρέπει να πληρώσουν γι' αυτό. Ούτε αυτοί είναι καλά παραδείγματα καλής διαχείρισης για άλλες χώρες. Γι' αυτό αν δεν βάλουμε κριτήρια όπως ποιοτικά κριτήρια ανισότητες στο εισόδημα, έρευνα και παραγωγικότητα της ενέργειας, ξεγελιόμαστε. Λέτε ανταγωνιστικότητα. Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά τι κάνει μια οικονομία ανταγωνιστική, μόνο τερ, μέσω του εργασιακού, 20% είναι τα, τα εργατικά. Αν δεν δούμε την ενέργεια, την παραγωγικότητα μέσω της έρευνας, ξεγελάμε τους εαυτούς μας. Δέστε πόσο ε, ευάλωτοι είναι οι Ιαπωνέζοι στη βιομηχανία τους. Δέστε. Έγιναν μια από τις πιο ευάλωτες κοινωνίες στη γη. Για το ιδιωτικό χρέος δεν λέει τίποτα το κείμενο και όμως ξέρουμε ότι αυτό δημιουργεί πολλές ανισορροπίες. Και μετά διάφορες επιπτώσεις δευτερογενής. Και να δούμε συστημικές αντιδράσεις Πάμε χάρη τα πλεονάσματα μερικών χωρών εξορισμού είναι ελλείμματα άλλων. Αν θέλουμε να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα πρέπει να δούμε και το άλλο σκέλος. Γιατί η γη στο σύνολό τη δεν βγάζει πλεόνασμα. Ποιο θα απορροφήσει το, το, το πλεόνασμα αυτό για να δημιουργήσει έλλειμμα. Οι αριανοί, οι μικροί πράσινοι, τα μικρά πράσινα όντα. Είμαστε κι εμεί πράσινοι αλλά δεν το κάνουμε αυτό κυρώσεις και ποινές, μην μου λέτε γι' αυτά, αν δεν μιλάτε και για κίνητρα. Ε, οι Γερμανοί βλέπουν τις ε, κυρώσεις σαν κίνητρα. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι μια αντίληψη που αφορά μόνο τους Γερμανούς, δεν συμφωνεί με την πραγματικότητα. Είναι σημαντικό αυτό το νομοθέτημα για να έχουμε οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη. Αλλά είτε μας αρέσει είτε όχι πρέπει να συνδεθεί με δύο άλλες βασικές παραμέτρους που δεν συζητιόνται εδώ και τις ξαναείπα. Είναι οι εξή. Πρώτον, μια συνολική φορολογική πολιτική. Μερικοί από εμάς θεωρούμε ότι πληρώνουμε πολύ φόρο, αλλά μερικοί άλλοι δεν πληρώνουν πολλά και πρέπει να φροντίσουμε να πληρώνουν και αυτοί. Αν θέλουμε να πουλήσουμε το πακέτο αυτό στους πολίτες μας, θα πρέπει να προχωράμε με την ίδια ταχύτητα και στο άλλο μέτωπο για τα φορολογικά. Και το δεύτερο που λείπει είναι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος. Πολλά έχουν γίνει, αλλά για τα δεσμευτικά νομοθετήματα, μην μιλάμε τώρα για υποπτίες και τέτοια, αποφασίσαμε να έχουμε νέους αστιφύλακες στα θέματα εποπτείας. Οι κανόνες όμως δεν άλλαξαν και πρέπει να αλλάξουν. Και βλέπουμε μεγάλη αντίσταση να μην αλλάξουν. Έχουμε μεγάλες τράπεζες που συμπεριφέρθηκαν ανεύθυνα. Πρέπει να πληρώσουν την ανευθυνότητά τους. Και αν οι πολίτες δεν τα δούνε αυτά, να κινούμαστε με την ίδια ταχύτητα στις αλλαγές όπως κάνουμε σε αυτό εδώ το θέμα, πάλι θα αισθανθούν ότι πάμε να τους ξεγελάσουμε. Ξεγελάσουμε και δεν θα τον ανεχτούν. Η Κορίν άνοιξε τη συζήτηση. Είχαμε μια διμερή συζάτηση, συνάντηση. Καλή αυτή η μέθοδος εργασίας. Θα έχουμε φαντάζομαι μερικές εβδομάδες έντονης συζήτησης και συνεργασίας. Πρόεδρος Φίλιπ Σόφισα, παραπάνω χρόνο επειδή είσαι ο μόνος πράσινος ομιλητής, να ξέρετε ότι γι' αυτό εξηγεί το γιατί σου άφησε να μιλήσεις τόση ώρα. Δεν ισχύει για τους άλλους. Και κατεβαίνω και ο κουρτίνες για να μπορώ να σας βλέπω καλύτερα. Γιατί με θαμπώνει ο ήλιος. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι και εγώ πολιτικός εδώ και κάμποσα χρόνια και βλέπω τις διαφορές στις χώρες μας συνήθως η, η κυβέρνηση θεωρεί την αντιπολίτευση ως μέρος του προβλήματος και η αντιπολίτευση αντίστροφα το ίδιο ως προς την κυβέρνηση. Άκουσα τον κύριο Μπούλμαν, άκουσα να μιλάει για έξυπνα και λιγότερο έξυπνα σύμφωνα κλπ. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία σχετικά με το περιθώριο ελιγμών στην κυβέρνηση. Και εγώ έχω κάνει υπουργό. Και μπορώ να πω με σιγουριά, κατά τη γνώμη μου, οι κυβερνήσεις προσπαθούν όσο μπορούν να ξεφύγουν από τις ευθύνε του. Καμιά κυβέρνηση δεν θα πάει για εκλογές έχοντας, κάνει, έχοντας πάρει αποφάσεις που δεν αρέσουν στο εκλογικό σώμα. Και οι περισσότερε από τις αποφάσεις αυτές έχουν σχέση με τις δαπάνες. Πριν τις εκλογές όλες οι κυβερνήσεις, είτε αριστερές, είτε κεντρό, είτε δεξιές, πριν τις εκλογές ο καθένας θέλει να ξοδεύει. Δυστυχώς όμως ο εκλογικός κύκλος δεν συμπίπτει με τον οικονομικό κύκλο. Μερικές φορές είναι καλά τα μέτρα αυτά, τις περισσότερες φορές δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Σε μερικές από τις προτάσεις που έχω υποβάλει για τις εκθέσεις αυτές σας καλώ να δούμε αν το να μιλάμε για ένα βλακώδες σύμφωνο και άκαμπτο αληθεύει. Πρέπει να σκεφτόμαστε ως ευρωπαίοι πολιτική, και όχι ως εθνική πολιτική. Δύσκολο πράγμα αυτό. Αν δεν υπάρχει πίεση εκ των έξω για πειθαρχία στις κυβερνήσεις που έχουν την πολιτική ανάγκη ή πίεση να αυξήσουν τις κρατικές δαπάνες, άρα να επιβαρύνουν την οικονομία τους και την οικονομία άλλων χωρών, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο αυστηροί με κυρώσεις για την πειθαρχία. Δεν με ενδιαφέρει να εφαρμόσουμε τις κυρώσεις, αλλά αν κανένας δεν σε επιβλέπει και οι εκλογείς λένε δώσ' τα όλα, τότε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να πατήσουμε το φρένο για να ισχύσει αυτή η μακροοικονομική πειθαρχία που απαιτείται. Ευχαριστώ. Λίο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η δημοσιονομική πλαισίωση των χωρών ε, μελών είναι το, πιο, είναι το λιγότερο ευαίσθητο μάλλον ε, κομμάτι του πακέτου. Η κυρία Φόρτ έκανε, επετέλεσε τεράστιο έργο για να, μιλήσει για, τη, για να καταφέρει να πετύχει σύγκληση των πολιτικών ομάδων, ιδιαίτερα για τα πιο τεχνικά ζητήματα. Την ευχαριστώ. Μάλιστα με καθησυχάζει και όσον αφορά τη θέση της Επιτροπής για την χρήση του ορισμού των κατάλληλων ε, μέσων προβολής. Παρ' όλα αυτά παραμένουν ε, ε, πράγματα με τα οποία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, παρόλο που είμαι σίγουρος ότι έχουν ε, μεγάλη καλή θέληση όλοι. Εμείς λοιπόν προτείνουμε να απομονωθούν οι δημόσιες επενδύσεις στους εθνικούς λογαριασμούς. Κατάλαβα ότι την ίδια άποψη συμμερίζονται και ορισμένοι από το ΕΛΚΟ, όπως ο κύριος Καρσία Μαργάγιο. Χαίρομαι γι' αυτό, αλλά άλλοι συναδελφοί του δεν συμφωνούν. Δεύτερον, ε, το να είναι πιο σοβαρές οι κυρώσεις. Δεν με εκπλήσει, μια από αυτήν η πρόταση που έρχεται από τους φιλελεύθερους και δημοκρατικούς. Η τροπολογία όμως 183 του κύριου Λάμπερτς που πάει προς την ίδια κατεύθυνση, αυτή με εκπλήσει. Σου υπενθυμίζω αγαπητέ Φιλίπ ότι η ίδια η αρχή του αυτοματισμού των κυρώσεων φέρνει, δυσκολεύει μάλλον την δυνατότητα των αντικυκλικών πολιτικών που βοήθησαν να βγει η Ευρώπη από την κρίση και να σωθεί ο κόσμος από την καταστροφή. Η συζήτηση αυτή μου φαίνεται ζωτική σημασίας. Πολλοί σήμερα λένε να βγούμε από τα πυρηνικά, ναι, αλλά πώς θα χρηματοδοτηθεί κάτι τέτοιο αν δεν μπορούν οι χώρες ε, να χρεώνονται γι' αυτό. Πολλοί συνάδελφοι τώρα μέσω των τροπολογιών τους εκφράζουν την ε, θέλησή τους να μην θέλουν τα κράτη-μέλη να υποφελούνται από δυνατότητες απόκλησης, εξαιρέσεων. Ναι, εντάξει Φιλίπ, έτσι κι αλλιώς ε, η αγορά απέτυχε, πολλές τράπεζες απέτυχαν, αλλά χωρίς τέτοια μέτρα πολλές τράπεζες δεν θα υπήρχαν σήμερα. Θα κινδύνευε η ίδια η Ευρώπη, οπότε άμα θέλεις να τα συζητήσουμε. Αλλά είμαι ιδιαίτερα επικριτικό για τροπολογίε πολλών συναδέρφων. Τέλο, για την ex post αξιολόγηση. Αναφέρθηκε σε αυτήν η Βίκη πριν από λίγο αξιολόγηση των κανόνων ex post. Πιστεύω ότι πέρα από τους ποσοτικούς δείκτες θέλουμε και ε, μια ποιοτική αξιολόγηση. Σήμερα γίνεται συζήτηση για τους δείκτες πλούτου. Οι οικολόγοι φίλοι θα τα ξέρουν. Εμείς θέλουμε να αξιολογούνται όλες οι πολιτικές, ιδιαίτερα όταν υποστηρίζουν ότι βοηθούν την ανάπτυξη μέσω φοροαπαλλαγών. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει συμβιβασμό. Είμαι στη διάθεση και τη κυρία Φόρτ και όλων των σχεδόν εισηγητών για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Από όσο όμως έχω ακούσει μέχρι τώρα, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός για ε, το τελικό αποτέλεσμα όσον αφορά αυτό το πακέτο οικονομικής ε, διακυβέρνησης. Γιώργαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ αυτό που είπε η Σιλβί Ότι θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις χώρες, όχι μόνο ο καθένας στη χώρα του. Και θα ήθελα να πω από την προοπτική αυτή ότι στην ομάδα μου υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εξετάζουν ε, κριτικά αυτά που προετοιμάζουμε και έχουν πολλές κριτικές να παρουσιάσουν. Η κριτική αυτή βασίζεται σε αυτά που είπε ο Φίλιπ Λαμπέρ αλλά και ο Γιάννη, δηλαδή ότι οι τράπεζες είναι εκείνες οι οποίες οδήγησαν στην χρέωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένε χώρες ε, είχαν κακή οικονομική πολιτική, αλλά η κύρια ευθύνη βρίσκεται στις τράπεζες. Και γι' αυτό θα ήμασταν εμείς κατά του να υπάρξει τώρα μια δέσμη νομοθετική που έχει σαν στόχο η ευθύνη αυτή της υπερβολικής χρέωση να μεταφερθεί στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το δεχτούμε. Γι' αυτό υποβάλαμε και κάποιες τροπολογίες οι οποίε ε, προ όψε δεν δίνουν την έμπαση γλωσσική μορφή, αλλά πάνε πολύ πιο μακριά, παραδείγματο χάρη, το θέμα τη εποπτεία. Θέλουμε να το αντικαταστήσουμε από συντονισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμεί δεν είμαστε καθόλου ενάντια σε μια λογική, σε ένα λογικό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών τη ενωση ε, Και άλλο αυτό και άλλο όμω η εποπτεία, γιατί το υπάρχει ενα υποπτη και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι υποκεινται στην ε, εποπτεία αυτή. Ενώ ο πολύ καλύτερο είναι ένα συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χαρών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το δημοσιονικό δίκαιο πλήττεται εδώ που είναι ένα βασικό δικαίωμα των εθνικών κοινοβουλίων. Εδώ δεν μπορούμε να παρέμβουμε, θα πρέπει αυτό να εξακολουθεί να τη χάνει σεβασμό. Και έτσι το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο επί ίσης όρης όλων. Αυτό σημαίνει ότι όσον αφορά και τις κυρώσεις εμείς δεν είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιώδεις για τις ε, προτάσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής. Εάν τελικά όμως όπως προβλέπετε επιβληθούν, ε, προβληθούν μάλλον καιρώσει, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι διαφανείς και θα ακολουθούν ε, τις αρχές του κράτους δικαίου. Γιατί κάποια που λέγονται εδώ ότι πρόκειται να γνωθούν και κλεισμένων των θερών κλπ. Αυτά δεν θα ήταν καθόλου διαφανή. Αν υπάρχουν λοιπόν καιρώσεις θα πρέπει να ακολουθήσουμε αρχέ κράτου δικαίου. Όσον αφορά τι ανισορροπίε, ελέγξαν διάφορα και θα ήθελα να τα τονίσω. Δεν αρκεί δηλαδή να αναφερόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη χώρα και να πούμε μία συγκεκριμένη χώρα έχει έλλειμμα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και μία ιστορική αγορά. Και η ιστορική αγορά έχει ανισορροπίε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τη συνεργασία των διαφόρων ε, εθνικών οικονομιών και ελέγχθη είδο ότι όπου υπάρχει ένα έλλειμμα υπάρχει από την άλλη μεριά ένα πλεόνασμα. Αυτά σχετίζονται μεταξύ του και θα πρέπει να τα δούμε πώς συσχετίζονται ακριβώς. Όσον αφορά το βαθμολόγιο, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε η συνάδελφο Δανούτα Χίπνερ. Εμείς θα θέλαμε τελικά να αναφέρετε κάτι στην ε, νομοθετική δέσμη. Αλλιώς φοβούμεθα ότι όπως έγινε και με την Ελλάδα θα χρησιμοποιείται αυτό μόνο για να μπορούν συγκεκριμένες χώρες με την αρχή της κατονομάζω ε, και τροπιάζω να αναφέρονται αυτές οι χώρες ε, στα ΜΜΕ κλπ. Αυτές οι εκστρατείες όμως ε, του κατονομάζω και τροπιάζω δεν είναι πολύ χρήσιμες γιατί είδα τι έγινε στη Γερμανία με την Ελλάδα γιατί δεν μπορεί κανένας να πει Ελλάδα σήμερα στη Γερμανία για να μην ρηχτούν όλοι και να αρχίσουν να λένε ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτό δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί στο, στο μέλλον. Δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτού του είδους τις διαδικασίες στο μέλλον. Και τέλος, θα ήθελα να τονίσω το εξή. Ε, δεν θέλω να πω ότι, κανένας ε, δεν, ε, ότι κάποιοι δεν έχουν εργαστεί σωστά στην Κομισιόν. Ε, όχι, όχι. Απ' την άλλη μεριά όμως στην νομοθετική αυτή δέσμη η Κομισιόν βρίσκεται κάπως υπεράνω όλων των πραγμάτων σαν να απομηχανής θεός προτείνει κάποια μέτρα, προτείνει κάποιες κυρώσεις χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθεί και να αιτιολογήσει τίποτα. Ε, λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει και η Κομισιόν ε, να παρουσιάσει ανοιχτά τα χαρτιά της ε, αυτό που θέλουμε είναι ότι θα πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε της η Κομισιόν και θα πρέπει αυτό που προτείνει να το προασπίζει και δημόσια. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Και τότε θα συμφωνούσαμε. Αυτό για μας είναι αυτό το σημείο. Νομίζω ότι ώρα ξεπέρασα το χρόνο γόρευσής μου και σταματάω εδώ. Thank you very much. Uh, next, Edward. Ευχαριστούμε, Edward. Θα μιλήσω πάνω στην έκθεση ΦΕΙΑ περισσότερο και όχι τόσο για την έκθεση της Σιλβή. Γιατί ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τα ευρωμόλογα, συμφωνούμε. και τις τροπολογίες μου και τις προτάσεις μου στην έκθεση ΦΕΙΟ θα τους έβαζα ως τίτλο «Μην ε, μαστιγώνετε το άλογο». Ίσως, αυτό το λέω για τις κυρώσεις, γιατί όταν θέλετε να επιβάλλετε τις κυρώσεις, το θέμα είναι να βοηθήσετε τη χώρα να μπει στο αυλάκι, να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Οπότε πρέπει να είμαστε μάλλον μετριοπαθείς. Καλύτερα να είμαστε μετριοπαθείς και να έχουμε τέτοιες ε, κυρώσεις που όμως να τις εφαρμόζουμε αποτελεσματικά παρά να έχουμε υπερβολικές κυρώσεις προβλέψει και όταν έρθει η ώρα της εφαρμογής τους να διαπιστώσουμε ότι δεν γίνεται. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να εισάγουμε κάποια ελαστικότητα. Εξαρτάται κάθε φορά από την οικονομική κατάσταση απέναντι στην οποία βρισκόμαστε. Γιατί κάποιες χώρες μπορούν να πληρώσουν τι κυρώσει, άλλε χώρες ίσως να είναι σε τόσο ε, απελπιστική κατάσταση που να μην μπορούν. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και ε, κυκλικά μέτρα διόρθωσης ανάλογα με το ΑΕΠ. Στο θέμα τώρα της ε, ευθύνη μπορούμε να συμφωνήσουμε εφόσον έχουμε πραγματικά εναρμονισμένο χώρο. Ε, έχει μετρηθεί καλά, έχει συμφωνηθεί από όλου. Και χωρίς να καταδεικνύουμε κανέναν για το θέμα των δημοσίων δαπανών. Γιατί όλες οι δημόσιες δαπάνες, είτε πρόκειται για συντάξεις, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο, ακόμα και το ιδιωτικό χρέος, αποτελεί ένα βάρος στο θέμα του contingency liability. Συνεπώς, πιστεύω και πρέπει να μελετήσω το σχετικό συμβασμό, ίσως τελικά καταφέρουμε να συμφωνήσουμε εφόσον διαπιστώσουμε ότι τηρούνται τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να γίνεται και σύνδεση με την απασχόληση και την ε, αηφόρο ανάπτυξη στην πραγματικότητα. Το τελικό δηλαδή αποτέλεσμα, αν δείτε τις προτάσεις μας, πρέπει να είναι τέτοιο που να λέμε ότι θα καταλήξουμε σε περισσότερη απασχόληση μετά την ανάκαμψη από την ε, κρίση. Γιατί θα έχει φροντίσει σε αυτό η νομοθεσία μας. Η εποπτεία τώρα πρέπει να χαίρει διαφάνειας. Και όταν ε, λέμε ότι τα κράτη-μέλη λογοδοτούν στο Κοινοβούλιο, πρέπει να τους ζητάμε να έρχονται και να μας εξηγούν ποια είναι η κατάσταση και να έχουν και το δικαίωμα να ζητήσουν να έρθουν και να μας εξηγήσουν, χωρίς να τους το έχουμε ζητήσει εμείς αυτό. Όσον αφορά τώρα το βαθμολόγιο, είναι, πώς θα το πω, ενδιαφέρον ότι στην αρχή ήμασταν κατά του να ε, τα βάζουμε με τον έναν ή τον άλλον δείχτη, λέγαμε ότι θα έπρεπε να είναι ελαστικοί οι δείκτες του βαθμολογίου και από την άλλη μεριά ερχόμαστε και μιλάμε για άλλες συμφωνίες όπου οι δείκτες κατονομάζονται και συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί να υπάρχει εξαίρεση εδώ. Να υπάρχουν και να πούμε ότι είναι και ανοιχτή, ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλοι δείκτε. Στο κατά κατω υπάρχουν και ορισμένοι που είναι ζωτική σημασία. Γιατί να μην του έχουμε συμπεριλάβει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τόφμαν. Äh, Ευχαριστώ, Βράδυ. Είμαι σκιώδη για την ε, ε, ομάδα μου της έκθεσης και θα περιορίσω τις παρατηρήσεις μου σε αυτό. Όσον αφορά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, νομίζω ότι εφαρμόσουμε τώρα ένα νέο σύστημα που δεν γνωρίζουμε καθόλου μέχρι στιγμής και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε σωστά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε εκείνο το σύστημα το οποίο πραγματικά συμβάλλει στην ανείχνευση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Τίποτα περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Και δεν πρέπει να ανακαλύψουμε τους καλούς και τους κακούς ή να ε, ε δίρουμε, αν μπορώ να το πω έτσι, κάποιες χώρες. Τουναντίον, Εάν υπάρχει ε, μια μακροοικονομική ανισορροπία και διορθωθεί έγκαιρα, αυτό δεν είναι μόνο προστασία για τις άλλες χώρες, αλλά προστασία και για την ίδια τη χώρα. Αν έγκαιρα είχαμε κατανοήσει τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στην Ελλαδία και είχαμε δράσει έγκαιρα, τότε δεν θα είχαν προστατευτεί μόνο οι άλλες χώρες, αλλά ιδίως η Ελλάδα ή η Ιρλανδία. Θα είχαν αποφύγει πολλά γιατί εκείνες υποφέρουν περισσότερο. Και έτσι θα πρέπει να εξτάσουμε και τον βαθμολογικό πίνακα. Και νομίζω ότι αυτός ο πίνακας θα πρέπει να είναι ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης, όπως το προέβλεψε και η Κομισιόν. Και θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε αυτό το βαθμολογικό πίνακα από εκείνο που θα έχουμε μετά, από το σχέδιο δηλαδή εξυγίενσης που θα πρέπει να λαμβάνει συνεχώς υπόψη τις αρχές της Ατζένας 2020. Αλλιώς ε, δεν είχε κανένα νόημα η Ατζέντα 2020, αλλά το βαθμολόγιο, ο βαθμολογικός πίνακας δεν επιτρέπεται να αναμειγνύει την ανείγνευση των μακροεκοπικών ισορροπιών και ένα ενδεχόμενο μελλοντικό μοντέλο που θέλουμε να καθίξουμε με την Ατζέντα 2020. Δύο πράγματα ακόμα. Αυτό που φαίνεται θα πρέπει να συζητήσουμε προσεκτικά και χαίρομαι που συζητιέται αυτό θετικά μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ποια είναι, ποιος είναι ο ρόλος της, ε, του Κοινοβουλίου, γιατί η Κομισιόν προβλέπει πολύ μικρό, για να μπω κανένα ρόλο για το Κοινοβούλιο. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να παρεμβαίνει στι εκτελεστικές εργασίε στο Κοινοβούλιο, αλλά από την άλλη μεριά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλαμβάνει οπωσδήποτε τι πολιτικέ του ευθύνε. Και θα πρέπει να δούμε και ποιο είναι ο ρόλο τη Κομισιόν. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει ένα πολύ ισχυρό ρόλο. Θεωρώ ότι η Κομισιόν θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο στο μηχανισμό αυτό και γι' αυτό στην ε, ομάδα μου προβλέπω μία σειρά ε, ψηφοφοριών αντιστραμμένης ειδικής πλειοψηφίας, γιατί έτσι μπορούμε νομίζω να βελτιώσουμε τον ρόλο της Κομισιόν. Τέλος, όσον αφορά τις συμμετρικές ε, εποπτείες όπως πρότεινε ο συνάδελφος Πλάμπρης προηγουμένως. Βέβαια εντάξει, ο φατμολογικός πίνακας πρέπει να είναι συμμετρικός. Ε, δηλαδή μπορεί να έχει η, από τη μια μεριά να υπάρχει ένα υπερβολικό εξωτερικό έλλειμμα και με φορά να υπάρχει ένα υψηλό εξωτερικό πλεόνασμα. Αλλά ξεκινώντα από εκεί να πούμε ότι αν έχει μια χώρα ένα πρόβλημα να δούμε τι έχει γίνει με τις άλλες χώρες, τι γίνεται, δηλαδή εάν μια χώρα όπως η Ιρλανδία έχει χαμηλούς φόρους ή μια χώρα όπως η Ισπανία που δίνει πολύ τεράστια ε, κίνητρα για επενδύσεις, εάν έχουν δημιουργηθεί έτσι κάποια κίνητρα και μετά λέμε σε μια εταιρεία ότι εσύ φταίς γιατί πήγες στην Ισπανία και επένδυσες εκεί, αυτό είναι προβληματικό. Θα πρέπει λοιπόν νομίζω να δούμε τα πράγματα προσεκτικά και να διαφοροποιήσουμε όσον αφορά την κατανομή αυτή του άχθους της ευθύνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Very much. Uh, now we come to... Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε στον κύριο Χόκμαρκ. θα χρειαστεί να φύγω για λίγο το πρόεδριο. Αν ε, ε, δεν γυρίσω μέχρι να τελειώσει, η επόμενη μιλήτρια είναι η Ευχαριστώ. Λέω ο κύριος Χιάκμαρ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Υπάρχουν πολλά θέματα για τα οποία συμφωνούμε. Από την μεριά όμως νομίζω ότι χάσαμε λίγο την αίσθηση του επίγοντος συζητώντας τα εδώ. δεν έχει περάσει και πολύ καιρό που έζησαν μεγάλη κρίση και ζουν κάπου στις χώρες μας που αφορά και τη δική του σταθερότητα και την κοινή σταθερότητα και όταν συζητάμε δαπάνες μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και ανεργία ε, όταν βρισκόμαστε παγιδευμένοι μέσα στην κρίση, όπου πάμε όλο και πιο βαθιά, και όταν συζητάμε πώς θα γίνει η ανάκαμψη, αν νομίζουμε ότι αυτό θα γίνει μόνο με δαπάνη και με ελλείμματα, έχοντας τις εμπειρίες που έχουμε ζήσει, τότε δεν μάθαμε αυτά που θα έπρεπε να έχουμε μάθει. Και όταν συζητάμε τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον, δεν είναι δυνατόν να πάρουμε όλα αυτά μαζί υπόψη. Γι' αυτό πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Έχουμε την τάση να συζητάμε ποιες είναι οι σωστές πολιτικές για το μέλλον. Πολύ δύσκολο αυτό να οριστεί. Είναι σαν να ψάχνουμε να βρούμε το Άγιο Δισκοπότηρο. Γιατί συζητάμε εδώ. Να αποφύγουμε τα λάθη που μας οδήγησαν να μπούμε στην κρίση επιτρέποντας μεγάλα χρέη μεγάλα βάρη. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και όταν συζητάμε για κυρώσεις, έχει σημασία αυτό. Διότι η ευρεία εποπτεία των οικονομικών πολιτικών καθιστά δύσκολες τις κυρώσεις. Γιατί μετά θα έχουμε αυθαίρετες συζητήσεις τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στην οικονομική πολιτική. Γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε για το βαθμολόγιο το scoreboard διότι αν το επεκτείνουμε το scoreboard και τον σύμφωνο σταθερότητας το κάνουμε το σύμφωνο εποπτείας της οικονομικής πολιτικής δεν θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τις εμπειρίες της κρίσης όσο πιο στενά είμαστε εστιασμένοι στους κανόνες που χρειάζονται για την οικονομική βιωσιμότητα, έλλειμμα, έλλειμμα τριχουσών συναλλαγών, για τους μεσοπρόθεσμους στόχους, κυρώσεις που, που να τους όλοι, διότι αν πάμε να τα κάνουμε όλα μαζί δεν πετύχουμε τίποτα. Αν εστιάσουμε την προσοχή μας στα σημαντικά, τότε το σύμφωνο σταθερότητας θα λειτουργεί και μετά μπορούμε να συζητήσουμε ποια είναι η σωστή οικονομική πολιτική στο μέλλον. Πρώτα πρώτα πρέπει να έχουμε σταθερότητα. Ευχαριστώ. Περβάνς. Ευχαριστώ. Τρία πράγματα. Φυσικά θα συζητήσουμε, φυσικά το Συμβούλιο θέλει να κλείσει μέχρι τον Ιούνιο. Πολλά συζητιόνται στο Συμβούλιο, το Ευρώ, στο Ευρωγκρουπ. και έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε λίγο, το χρέος, το ύψος του χρέους, τη διάρκεια κλπ. Στο μεταξύ έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και άλλα έγγραφα. Στην αρχή, πριν από καιρό, η κυρία Βόρτμαν Κόλ μας είπε να μείνουμε σε έξι κείμενα μόνο. Πάνε αυτά. Υπάρχουν στρατηγικές οικονομικής πολιτικής που αρχίζουν και εφαρμόζονται που αγνούν εντελώς τα κείμενα αυτά. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να εκπέμψουμε ένα έντονο πολιτικό σινιάλο. Ο πρόεδρος Τρισέ χθες πήρε θέσεις Πήρε θέση μάλλον ως προς το πακέτο αυτό. Εγώ έρχομαι από τη Γενέβη όπου συναντήσαμε τον πρόεδρο Σαμαγιάλ, τον πρόεδρο του ΟΗΤΕ και παραξενεύεται πως τόσες κεντρικές τράπεζες, ιδιωτικές τράπεζες κάνουν έρευνες για το θέμα της αγοράς εργασίας και δεν ανησυχούν για το πώς οι ίδιες οι τράπεζες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Θυμάμαι δε αυτά που μας είπε ο Ζακ Ντελόρ την περασμένη Δευτέρα και για την κοινωτική μέθοδο και για τον τελείως άχρηστο χαρακτήρα ο κύριος Κρούκμαν, βραβείο Νόμπελ, το αμφισβήτησε για το μοναδιαίο κόστος εργασίας και το πόσο μετράει την ανταγωνιστικότητα. Στο ΟΗΤΕ το ίδιο πράγματα μας είπανε. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο να σας τα αναλύσω αυτά. Ας σκεφτούμε τι κάνουμε εδώ. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Μερικοί λένε ότι αυξήθηκαν υπερβολικά οι μισθοί σε μερικές χώρες του Νότου. Να το καταδικάσουμε. Να το διορθώσουμε. Η ανάλυση του πώς λειτουργούν αυτές οι οικονομίες μας δείχνει ότι αν παρέκλειναν στην αρχή οι μισθοί ήταν γιατί υπήρχαν πληθωριστικές προσδοκίες οι οποίες μετά διορθώθηκαν αλλά η αύξηση των τιμών οφείλεται σε δυσλειτουργία της αγοράς των προϊόντων και όχι των μισθών. Τεράστιες παρανοήσεις κάνουμε δηλαδή. Δεύτερο, ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που θα επανέλθω σε κάτι. Εγώ δεν έχω καταθέσει καμία τροπολογία για τα έξι κείμενα. Για τον εξής απλό λόγο. Ως μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης Κοινωνικά Θέματα ήμουν εισηγήτρια για τρεις γνωμοδοτήσεις από τις έξι. Ξέρω ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα στην δική σας επιτροπή όλοι, όλοι οι συμβασμοί γίνονται. Εγώ σας ζητάω, ζητάω να λάβετε υπόψη σας τι ψηφίσαμε στην Επιτροπή Απασχόληση Κοινωνικά Θέματα. Γιατί αν θέλουμε να βγούμε από το Λούκι και να αρχίσουμε να περπατάμε όρθιοι στα πόδια μας, πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ψηφίστηκε και αλλού. Και δύο-τρία άλλα σημεία από την Επιτροπή Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την έκθεση της κυρίας Βόρτμαν Κόλ προτείνεται ένα εναλλακτικό κείμενο σχετικά με το Prudent Fiscal Policy που κανένας δεν μπορεί να την ορίσει. Εμείς ψηφίσαμε ένα συνθετικό κείμενο πιο καλό, κατά τη γνώμη μου, από το δικό σας. και μια δημοσιονομική πολιτική που θα είναι βιώσιμη και αποδοτική. Και το θέμα αυτό της βιωσιμότητας, μην το υποτιμούμε. Ε, δεν θέλουμε να κάνουμε ένα τεχνικό κείμενο κυρώσεων. Πρέπει να ορίσουμε ποια θα είναι η αυριανή οικονομική πολιτική και αν δεν μπει η διάσταση αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, θα παραμένουμε στο λάθος δρόμο. Για τις συντάξεις, κύριε Φεγιώ, ψηφίσαμε τροπολογίες που δέχονται αναφορά στις συντάξεις, αλλά ουδέτερα. Διότι μια οικονομική πολιτική της Ένωσης που δεν δέχεται να λάβει υπόψη τα στοιχεία του Golden Rule, πάμε χάρη για τις προκλήσεις του μέλλοντος, οι επενδύσει στην εκπαίδευση έχει προτεραιότητα. Σήμερα δεν έχουμε το δικαίωμα να το πούμε στο πακέτο αυτό. Πρέπει να το πούμε. Να πούμε ότι οι συντάξεις μέσω κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να τις δούμε με θετικό μάτι. Όχι, λέω εγώ. Όχι. Εγώ ζητάω τη βιωσιμότητα, την απόδοση του συστήματος των συντάξεων μέσω επιμερισμού. Για την έκθεση της κυρίας Βίκη Φόρντ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Η έκθεσή σας είναι σημαντική για κάτι που το συζητήσαμε στην Επιτροπή Απασχόλησης για το ότι αν όγι λέμε ότι να είμαστε καλοί Ευρωπαίοι ε, τότε ας φροντίσουμε να εξοπλιστούμε με τα εργαλεία για τη στρατηγική μας. Στην Ένωση έχω μία στρατηγική με την οποία εγώ δεν συμφωνούσα απόλυτα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Αν δεν έχουμε μία σαφή στρατηγική επενδύσεων, πάμε κόντρα στην στρατηγική αυτή. Δεύτερον, η Ένωση δεν είναι πολύ μεγάλη για να το κάνει όλα αυτά μόνη της. Αν δεν δει πώς οι δαπάνες των κρατών μελών συμβάλλουν στη στρατηγική αυτή, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Και αυτό πρέπει να μπει στην έκθεσή σας κυρία Φόρντ. Πολλά άλλα συζητήθηκαν στην Επιτροπή Απασχόλησης μην θεωρείτε ότι εσείς είστε έτοιμοι, ξεκίνησατε τους συμβασμούς σας συμπλην, συμπλην, και ότι θα ψηφίσετε. Γιατί υπάρχει μια διάσταση που την αγνοείτε και θα μπείτε σε μια στρατηγική που είναι στρατηγική των χαμένων. Μία τελευταία παρατήρηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Οι συντονιστέ τη Επιτροπή σα αποφάσισαν να υπάρχει μια έκθεση πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο και με ορίσατε υπεύθυνοι η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων, η Επιτροπή Προπολογισμών, σίγουρα και η Επιτροπή Απασχόλησης θα γνωμοδοτήσουν. Τόσο το καλύτερο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να είμαι το χεράκι κάποιου ο οποίος είναι αλλού και παίρνει αυτός τις αποφάσεις. Εγώ θέλω να δούμε στα έξι κείμενα που έχουμε μπροστά μας τι μπορεί να μπει σε ένα πακέτο που να λέγεται Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Γιατί εγώ δεν είμαι σκλάβος κανενός. Προς το συμφέρον του Κοινοβουλίου μας συμφέρει να έχουμε ένα ενιαίο κείμενο χωρίς ανακολουθίες έτσι ώστε να έχει λόγο ύπαρξης και το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί ξέρουμε ότι το Συμβούλιο δουλεύει όλο και περισσότερο με ανεξάρτητους συμπειρογνώμονες και ξέρουμε που μας οδηγούν αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Περβάνς. Ε, νομίζω ότι εκ της αρχής η πρόθεση της κυρίας ε, Τζονκό και των εισηγητών ήταν να ενταχθούμε στην στρατηγική 2020 Ξέρω εσύ δεν θέλετε το λόγο, αλλά έχω ακόμα δύο συνάδελφους που θα πρέπει να πάρω το λόγο. Εκτός αν είναι πάρα πολύ σύνομο αυτό που θέλετε να πείτε. Ναι, ήθελα να δώσω μια πληροφορία. Πολλά κάνουμε για να φροντίσουμε να εισακουστεί το κοινοβούλιο. Μαχηθήκαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Φανερόπαη που έγινε αυτό την περασμένη εβδομάδα και όλοι, και η Ελίζα κυρίω και όλοι, έχουμε αναφέρει ότι θέλουμε να εισακουστεί το κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεργαστούμε μαζί σου για το εξάμεινο, αλλά αυτό ήταν για να ενημερωθούν εκείνοι που δεν το ξέρουν ίσω. Με συγχωρείτε που διακόπτω τη συζήτηση, λέει κύριε Περές. Αλλά τότε δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να περάσει αυτό η δέσμη χωρίς να συμπεριλάβουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτό είναι που από την πρώτη αλληλεγγύη απόψε το έκανε απόλυτα σαφές κυρία Βαρτμακόλ. Να με δώσουμε το λόγο τώρα στου όλους δύο συναδέλφου του μπορείτε να επανέλθετε. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία στο θέμα της εποπτείας των ανισορροπιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα να το δούμε σωστά διαφοροποιημένο και με ακρίβεια. Δεν είναι καλό να είχαμε ένα σύστημα το οποίο δεν επιτρέπει σωστή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τους μισθούς, υπάρχει πολύ έντονη ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ίσως είναι αντιπαραγωγικό. δεν υπάρχει κανένα απόδειξη ότι η μισθή που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερη από τους άλλους των αντίων. Γιατί ε, πρέπει να έχουμε ισορροπία. Η, η καθορισμός των ε, συλλογικών συμβάσεων από τους ε, ε συλλογικούς εταίρους είναι η καλύτερη οδός για επίτευξη μιας ισορροπίας και γι' αυτό θα πρέπει αυτές τις συλλογικές συμβασίες να λαμβάνονται υπόψη όταν συζητάμε καλή κατανομή ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε επίδραση στην δημιουργία αυτών των μισθών και γι' αυτό ε, μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν σε τρία σημεία όσον αφορά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Καταρχήν θα πρέπει το εθνικό ε, πρότυπο του κοινωνικού διαλόγου να ληφθεί υπόψη. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε καλώς λειτουργούσες ε, δομές. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία δυνατότητα να επιβάλλουμε στην εθνική κυβέρνηση να αναμειχθεί στην ε, δημιουργία των μισθών. Θα πρέπει οι κυβερνήσεις να έχουν δυνατότητα να λάβουν υπόψη ε, την ελευθερία των εταίρων. Τρίτον, εάν υπάρχει ανάμειξη σε ένα διάλογο μεταξύ Βρυξελών και κρατών μελών, χωρίς να ληφθούν υπόψη ε, ε, οι κοινωνικοί εταίροι, θα μπορούσαν ίσως να υπάρχουν τεράστιες στρεβλώσεις. Για να λειτουργήσει κάτι στην πράξη θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά αυτές τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και που είστε και το λόγο, στον χρόνο. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, λέει ο κ. Έχω λίγες παρατηρήσεις. Καταρχήν προς τον φίλο Λιάμ. Καταρχήν, η αλλαγή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρηματοδοτεί στη Γερμανία από το ιδιωτικό τομέα και ξέρουμε γιατί. Δεύτερον, δεν πιστεύω ότι ε, μια, ε, ένας δημόσιος ε, πυρηνικός είναι καλύτερος από έναν ιδιωτικό. Όλα αυτά εξαρτώνται από την επιλογή που θα κάνει κανένας. Αυτή εδώ η δέσμη δεν έχει καμία σχέση με την αλλαγή από πυρηνική ενέργεια στι ανανεώσιμες πηγέ ενέργεια. Δεύτερον και επί του θέματος, θα ήταν σημαντικό νομίζω να παίρναμε λίγο χρόνο στην Επιτροπή, δεν ξέρω πότε, για να βγούμε από το σκεπτικό αυτό του εξετάζουμε μία-μία έκθεση και να εξετάσουμε από κοινού τις επιπτώσεις του συνόλου συμπεριλαμβανομένου και του Συμφώνου για το Ευρώ, τις έξι προτάσεις και το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τις, την κόκκινη γραμμή του, κανενός και, του καθενός συγγνώμη, και να κατανοήσουμε ποια είναι πραγματικά η άποψη ε, για κάθε θέμα. Όπως είπε και η κυρία Βόρτμαν Κόλ, θα συζητάμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και θα ξεχνάμε ότι το σύνολο πρέπει να εξεταστεί. Αυτή είναι μια ευθύνη που έχουμε όλοι εμείς δηλαδή. Μετά τις ψηφοφορίες θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σφάλαμε και τη δεύτερη φορά. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα προσπαθήσω να το συζητήσουμε αυτό και στους συντονιστές. Να σταματήσουμε δηλαδή ένα λεπτό, να βγούμε από το σκεπτικό αυτό, εξετάζουμε μία-μία-μία-μία έκθεση και νομίζω ότι η Κορίνη είπε ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε κάποιους συμβασμούς αν το συζητήσουμε το θέμα όπως σας προτείνω. Γιατί είχαμε κάποιες ανταλλαγές απόψε ακριβώς σήμερα το πρωί όπου είπαμε ότι ίσως για ορισμένα από τα θέματα συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες αλλά δεν είναι σωστό να τις αναφέρουμε εδώ. Ε, ε, ε, ορισμένοι φοβούνται αν δεν το κάνουμε στο πλαίσιο των έξι προτάσεων θα χαθούν οι πτυχές αυτές. Μπορούμε λοιπόν να βγούμε από αυτό το σκεπτικό του εξετάζουμε μία-μία τροπολογία, μία-μία έκθεση και να εξετάσουμε τη συνολική εικόνα. Ίσως θα μπορούμε να βρούμε κάποιο χρόνο να το κάνουμε αυτό. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πλήρης αίθουσα όταν το κάνουμε. Πρώτα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα πολλά να πω, αλλά θα δώσω το χρόνο μου στους συζητητές για να μπορέσουν να δευτερολογήσουν. Θέλω να τονίσω μόνο ότι πιστεύω ότι πολλά από τα θέματα που αναφέρονται σε διάφορες τροπολογίες και τις δικές μου και των συζητητών μας δίνουν τη δυνατότητα να ενώσουμε αυτές τις διάφορες προτάσεις. Θα παράσω σε ένα πρώτα, Κορίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους για τις παρατηρήσεις τους, για τα σχόλιά τους όσον αφορά την, το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου σταθερότητα. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια κοινή γραμμή. Είναι κρίμα που φεύγετε. Κρίμα. Κρίμα γιατί θα ήθελα να σχολιάσω το που βρισκόμαστε προς το παρόν. Γιατί και στον Οδομπάουμεν και σε άλλους Εξάλλου διαπιστώσαμε σήμερα ότι είμαστε και οι δύο επιστήμονες. Δεν μιλάμε μόνο για ένα ε, καλό σύμφωνο σταθερότητας και ένα τέτοιο σύμφωνο, και το λέω αυτό και για τον Κρίστιαν. Εδώ είμαστε μια οικονομική και νομισματική ένωση. Πρέπει να πάρουμε μαθήματα από την κρίση. Πρέπει να φροντίσουμε να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μόνο με το νομισματικό σκέλος. Άρα χρειάζεται ένα ευφιές πακέτο, ένα ευφιές σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Σφεν, μπορεί να λες να περιμένουμε. Μα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα από μόνο του αν εμείς δεν έχουμε τον ηγετικό ρόλο. Γιατί είναι και το είπαμε και το ξανάπαμε με τους εισηγητές ότι προκαλείται σύγχυση. Υπάρχει το πρόγραμμα σταθερότητας, υπάρχει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης για την ε, ε μακροχρονή εποπτεία, έχουμε τη στρατηγική 2020 και τώρα έχουμε και τους νέους αυτούς δείκτες ή τουλάχιστον παρουσιάζονται σαν νέοι στο πακέτο για το ευρώ. Σίγουρα μιλάμε για εποπτεία από τους ομότιμους, μιλάμε επίσης και για τεχνικά ε, σχέδια αναδιάρθρωσης. Πάντως εμείς και εγώ ως εισηγήτρια αυτό που θέλω είναι να πετύχουμε βιώσιμα δημοσιονομικά και βιώσιμη ανάπτυξη. Για μένα η προσέγγιση μου χρειάζονται και τα δύο. Η στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 περνάει ε, σε δεύτερο πλάνο, όπως έγινε και με τη στρατηγική της Λισαβόνας, γιατί τώρα οι επικεφαλής κατόχοι κυβερνήσεων ε, θα ασχοληθούν μόνο με τους ε, νέους δείκτες. Κύριε Μπερές, ξέρω ότι σας απασχολεί η απασχόληση, είσαστε πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης, αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο. Εσείς αναφερθήκατε σε πολλά θέματα που συμπεριλαμβάνονται στις τροπολογίες το κείμενο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο το προτείνω στην ε, έκθεσή μου. Χαίρομαι που κι εσείς συμφωνείτε και που το βάζετε κι εσείς στην έκθεσή σας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε προς μια κατεύθυνση που να ισχυριζόμαστε ότι είναι δικιά μας υπόθεση αυτός ο δρόμος. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης. Σήμερα μάλιστα ζήτησα από την Επιτροπή να φροντίσει να καθίσει μαζί μας, να ετοιμάσει ένα ε, πακέτο. Δεν είναι απ' έξω που θα μας έρθει. Εδώ, εμείς θα βάλουμε ό,τι θέλουμε στο πακέτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω να έρθει με καλές ιδέες. Αλλιώς θα το κάνουμε εμείς, γιατί θέλουμε μια έξυπνη προσέγγιση. Επί τότε θέλουμε να πετύχουμε τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Το Κοινοβούλιο το λέει στο ψήφισμα που εγκρίναμε πριν από μερικούς μήνες. Για να πετύχουμε τη στρατηγική αυτή, πρέπει να υπάρχει μια σαφής δέσμευση με στόχους και χρειάζονται και μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Εδώ συμφωνούμε. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε περισσότερο και να συζητήσουμε μετά πώς θα το πετύχουμε αυτό. Με κάποιες τροπολογίες ε, το είπα ποιο είναι το πρόβλημά μου, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε χέρι με χέρι και να προωθήσουμε το πακέτο αυτό. Ευχαριστώ. Δίκη. και εσείς. Περβάς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι χρειαζόμαστε απασχόληση και ανάπτυξη, αλλά δεν κολλάει στην έκθεση εδώ το πώς μπαίνει στον μηχανισμό. Είναι περισσότερο για την έκθεση της Κορίν που μιλάμε για τις οικονομικές πολιτικές. Δεν είμαστε συνεμοθέτες για την έκθεσή μου. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να ζητάμε πράγματα που μπορούμε να πετύχουμε. Τη διατύπωση που θέλεις μπορούμε να τη βάλουμε στην έκθεση της Κορίν κύριε Χαγνόη. Πολλές από τις τροπολογίες σας είναι λογικές, αλλά δεν σημαίνει ότι όλες θα μπουν στο συμβιβασμό. Κάποιες περιλαμβάνονται, αλλά για άλλες παλεύω ακόμα. Μπορούμε όμως να τις συζητήσουμε. Όμως, διαφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι η οδηγία που βελτιώνεται από το Συμβούλιο σε αυτήν εσείς διαγράφετε το θέμα της διαφάνειας. Το Συμβούλιο είπε ότι θα συμφωνήσει για τις υποχρεώσεις. Όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο για το πού πάνε τα χρήματα, για το πού είναι τα χρέη, όλα αυτά είναι θετικά. Οπότε διαφωνώ με μια προσέγγιση που λέει όχι, διαγράφεται η διαφάνεια. Όχι. Εκτός αν δεν σας κατάλαβα καλά. Ευχαριστώ. Η Ελίσσα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να δούμε λίγο τι είπαν οι συνάδελφοι. Πρέπει να δούμε το πακέτο αυτό ως μια απάντηση στα προβλήματα που έχουμε και αντιμετωπίζουμε. Έτσι πρέπει να το δούμε. Οι συνάδελφοι λοιπόν που απλώς θέλουν να μιλάνε για το πακέτο σταθερότητας και ανάπτυξης έτσι όπως έχει τώρα, είναι σαν να συμφωνούμε με την ιδέα ότι δεν λειτουργήσε. Μα γι' αυτό και προσπαθούμε να το αλλάξουμε το πακέτο, γι' αυτό προσπαθούμε το πακέτο αυτό να το κάνουμε καλύτερο. Γιατί ήταν μια μερική απάντηση. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία δεν καλύπτονται μόνο από το πακέτο σταθερότητας και ανάπτυξης. Για παράδειγμα, άρρητα στους στόχους, έλεγε 60% και 3% 3% ανάπτυξη της οικονομίας και πληθωρισμός 2%. Αυτό ήταν ολόκληρο το πακέτο. Αν προσπαθείτε να προβλέψετε 3% και 60% δεν είναι λύση για το πρόβλημα. Το πρόβλημα παραμένει και το πρόβλημα είναι έλλειψη αντικυκλικών δυνατοτήτων και η αντίσταση της Ευρωζώνης όταν υπάρχει κρίση, με τι μέσα, τι κάνουμε και οι αποκλίνουσες τάσεις μέσα στο ευρώ, χωρίς ικανοποιητική ανάπτυξη. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Τι θα κάνουμε, θα πάμε πίσω και θα πούμε στους πολίτες η λύση είναι κυρώσεις και μάλιστα πιο αυστηρές με απέτηση συμμόρφωσης. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε καλύτερα πώς μπορούμε να κάνουμε την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανθεκτικά και πιο σταθερά στοιχεία και πιο κατάλληλα για την καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Για να ολοκληρώσω πρέπει να εισαγάγουμε στοιχεία που επιτρέπουν σύγκληση και ανάπτυξη. Και αυτό δεν μπορεί να είναι μια διατύπωση καινή περιεχομένου. Αλλιώς θα είναι μια ευκαιρία που θα έχουμε χάσει. Και για να επανέλθω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Φέιο. Είπε γιατί 2020 για να επιστρέψουμε στο σωστό δρόμο, γιατί 0,5% ε, κάθε χρόνο για το έλλειμμα, πώς αυτά κολλάνε μεταξύ τους Μα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα προβλήματα είναι περίπλοκα και ότι είναι προτιμότερο να φροντίσουμε για αυτή την ε, αντίσταση και για την ε, εξυγίανση παρά να συνεχίσουμε να κάνουμε πολιτικά σφάλματα επιβάλλοντας υψηλές κυρώσεις και πολύ αυστηρούς κανόνες που τελικά κανένας δεν θα ακολουθήσει. Ή θα τους ακολουθήσουν μόνο μερικοί γιατί οι υπόλοιποι δεν θα τους εφαρμόσουν. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Άλλος εισηγητής. Τέσσερα λεπτά έχουμε ακόμα διερμηνία, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ, Σόφη. Θέλω να πω ότι χαίρομαι που μείνανε εδώ όσοι μείνανε. Ε, εδώ ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά μεταξύ μας, παρόλο που δεν έχουμε πολλούς μουσικούς. Ωραία, τελειώσαμε τότε στην ώρα μας και θα συνεχίσουμε.